Right, good, uh, Καλημέρα σα. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δυστυχώ ε, φτάνε τα τρένα. Ο πρόεδρο ε, Τρισέ είχε κλείσει να έρθει με ένα τρένο το οποίο ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν, ε, ακόμη και αν ο πρόεδρο τη ΕΚΤ δεν <laughs> είναι δυνατόν να κάνει ένα τρένο να λειτουργήσει όταν ακυρώνεται, αλλά χρειάστηκε λοιπόν πολύ χρόνο για να έρθει. Καταρχήν έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, να θεωρήσω ότι εγκρίνεται. Υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις, ε, καταρχήν. Έχουμε το workshop για την ε, οδηγία ε, για τον ε, νομοθεσία περί ασφάλειας. Ε, ξεκινά στις 10.30. Είναι στο 1G1, στο Αλτιέρο Σπινέλη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ δεν μπορώ να παρευρεθώ εκεί, γιατί θα πρέπει να παρευρεθώ σε ένα τριμερή διάλογο για την οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα για το short selling ε, θα σας δώσω μια ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο της 28 Ιουνίου. Η Κομισιόν παρουσίασε διάφορες προτάσεις ε, για συμβιβασμό που πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή και ο εισηγητής ζήτησε από την Κομισιόν να επανέλθει με νέα διατύπωση για ορισμένα άλλα ζητήματα και επίσης περιμένει ε, και feedback από το Συμβούλιο για ορισμένα από αυτά τα θέματα. Δεν ε, Επετεύχθη συμφωνία λοιπόν σε διάφορα κυρία ζητήματα σε ό,τι αφορά την απαγόρευση του CDS, την ε, δυνατότητα opt-in ε, και τη δυνατότητα opt-out και τις αστηρές προϋποθέσεις που απαιτεί η Επιτροπή ΕΚΟΝ ούτε συμφωνία σε σχέση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει ψηφοφορία στην Ολομέλεια του κειμένου που ήδη ψηφίστηκε στην ΕΚΟ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης ε, και να περάσουμε στο νομισματικό διάλογο με την ΕΚ. Το τελευταίο νομισματικός διάλογος με τον Πρόεδρο έλαβε χώρα στις 23 Μαρτίου και η επόμενη συνάντηση πιθανότατα θα λάβει χώρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Είχαμε λάβει και κάποια ενημερωτικά έγγραφα για την ε, δημοσιονομική λιτότητα και την ε, διαχείριση, τον αντίκτυπο ε, στα κράτη-μέλη, την αναδιάρθρωση του χρέους και τις συνέπειες στο ευρώ. Αυτά έχουν δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα και δυστυχώ λόγω πίεση του χρόνου δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε με τους εμπειρογνωμονε μας, αλλά φυσικά αυτό δεν μα σταματά από, το να θέσουμε ερωτήσεις για αυτού του τομεί. Και φυσικά έχετε ήδη λάβει τον κατάλογο των ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω εγώ να σας βοηθήσω το δυνατό περισσότερο στο να διασφαλίσω ότι ε, θα σεβαστούμε το χρόνο για τις ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι λαμβάνουν χώρα και άλλες συνεδριάσεις που τυχόν σε ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τρισέ, χαιρόμαστε πάντοτε που σας έχουμε εδώ, είναι ικανοποίησό μας ε, και συγγνώμη αν σας ε, πιέσαμε λίγο, τώρα έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Με χαρά βρίσκομαι ξανά στο Κοινοβούλιο και ενώπιον της ε, Επιτροπής σας ε, για μια τακτική ανταλλαγή απόψεων και μάλιστα σε μια στιγμή όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ε, σημαντικές αποφάσεις που εκκρεμούν ιδίως ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του νομοθετικού πακέτου της νομοθετικής διαδικασία για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω τι άκρονες προσπάθειες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με στόχο να προσεγγίσουν ε, λίγο τις απόψεις τους ό,τι αφορά το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Γνωρίζετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε στις 24 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κάνει μια χειρονομία καλή θέληση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχε ένα βασικό σημείο διαφωνία, η επέκταση τη αναστραμμένη δική πλειοψηφία στο προληπτικό σκέλο του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χρειάζεται η Ευρωζώνη επιγόντω ένα ενισχυμένο και φιλόδοξο πλαίσιο οικονομική διακυβέρνηση, διότι όπω δείχνει η σημερινή κρίση, αν χρειαστεί ε, κανείς ακόμη αποδείξεις γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές καταστροφικές απεπτήσεις ε, πολιτικές για τη δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών. Επομένως, χρειάζεται να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήταν, θα ήταν πάρα πολύ ε, καλοδεχούμενη μια τέτοια συμφωνία από τις παρουσες συνθηκες ουτως ώστε να καταστεί σαφες ότι θα αντλήσουμε τα διδάγματα από την κρίση. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Μετά την τελευταία μας συνεδρίαση που έγινε το Μάρτιο, έχουμε υιοθετήσει κάποιες κατευθύνσεις. Να σημειώσω, κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, ότι έχουμε την επόμενη συνάδριαση του Κοινικού Συμβουλίου σε 7 Ιουλίου και αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε λέω σε σχέση με την ε, μελλοντική νομισματική πολιτική δεν μπορεί να προδικάσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν ε, στις 7 Ιουλίου. με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μία όθηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη και περιμένουμε να συνεχίσει να αναπτύσσεται η παγκόσμια οικονομία αλλά και η εγχώρια ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα γιατί αυτός είναι και ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη οι τελευταίες ε, μακροοικονομικές ε, προβολές του προσυστήματος ε, ευθυγραμμίζονται με την εκτίμηση αυτή, διότι προβλέπουν ανάπτυξη μεταξύ 1,5 και 2,3% για το 2011 και μεταξύ 0,6 και 2,8% για το 2012. Κατά την άποψή μας, είναι ισορροπημένοι αρκετά οι κίνδυνοι ε, βέβαια σε ένα πλαίσιο μεγάλης ε, αβεβαιότητας. Ό,τι αφορά τις εξελίξεις των, ε, στις τιμές, βλέπουμε συνεχή όθηση των τιμών προς τα άνω, ιδίως στα πρώτα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη ήταν 2,7 το Μάιο και 2,8 βέβαια <clears throat> τον Απρίλιο. Στους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτός ο πληθωρισμός αφορά τις υψηλότερες τιμές ε, της ενέργειας ε, και των ε, αγαθών κοινή ωφέλειας. Ακριβώς λόγω των τιμών σε αυτούς τους τομείς αναμένεται ο πληθωρισμός να παραμείνει σαφώς πάνω από το 2% τους επόμενους μήνες. Τώρα, οι προβολές αυτές του Eurosystem που σας είπα δείχνουν ένα πληθωρισμό μεταξύ του 2,5 και 2,7 για το 2011 και μεταξύ του 1,1 και 2,3% για το 2012. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτά τα τρέχονται ψηλά ποσοστά πληθωρισμού να μην ε, μεταφραστούν σε ε, επιπτώσεις στο δεύτερο γύρο που θα είναι δηλαδή ψηλότερη ε, μέσω των υψηλότερων μισθών και της τιμολόγησης. Άρα να έχουμε πληθωριστικές πιέσεις ευρύτερες. Επίσης οι κίνδυνοι ε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών ε, αυξάνονται, σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη τις τιμές ενέργειας, ενδέχεται να έχουμε ταχύτερη αύξηση από την αναμενόμενη και ίσως χρειάζεται ε, να αυξηθούν ταχύτερα οι έμεση φόροι για να μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ γενικότερα στις τιμές θα ασκηθούν πιέσεις. Ό,τι αφορά την νομισματική ανάλυση, βλέπουμε ότι η νομισματική ανάκαμψη είναι σιγά σιγά πραγματικότητα. Βέβαια έχουμε αρκετά μεγάλη νομισματική ρευστότητα και έτσι μπορούμε κάπως ε, να απορροφήσουμε τις πιέσεις της τιμές. Ξέρετε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι προσδοκίες ό,τι αφορά τον, τον πληθωρισμό θα παραμείνουν ε, μέσα στα πλαίσια, μέσα στους στόχους μας που είναι να κρατάμε σε χαμηλά επίπεδα τον πληθωρισμό αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν ε, αυξήσαμε τα βασικά επιτόκια κατά 25 ε, ε, βασικές μονάδες τον Απρίλιο για να αντιμετωπίσουμε τη... τον κίνδυνο της αστάθειας στις τιμές αλλά δεν αλλάξαμε από τότε τα επιτόκια και όπως είπα και στην συνέντευξη τύπου την τελευταία που δώσαμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε κινδύνους ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών. Και βέβαια παραμένουμε σε επαγρύπνηση και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εγκαίρως και αποφασιστικά για να μην προκύψουν λόγω των τελευταίων εξελίξεων στις τιμές μεγαλύτερες, ευρύτερες, πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα. Επίσης αποφασίσαμε πρόσφατα να διατηρήσουμε τις ε, διαδικασίες διαγωνισμού με ε, σταθερή ε, τιμή. Και έτσι θα χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις μας μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2011. Ας έρθω τώρα στον τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Σε μια νομισματική ένωση η Κεντρική Τράπεζα όταν ε, ορίζει τα επιτόκια πρέπει να βλέπει τα πράγματα από ευρία οπτική γωνία. Το ίδιο ακριβώς ε, συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ, όπου δεν μπορεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον ΗΠΑ, ούτε και πρέπει άλλωστε να προσαρμόζει τα επιτοκιά της στις οικονομικές συνθήκες των τον ΗΠΑ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοούμε και την πολυμορφία, την ποικιλομορφία των δημοσιονομικών συνθήκων. Μετά την ε, δημοσιονομική κρίση όταν ξέσπασε, κρίναμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποια μη τυπικά μέτρα ώστε να υπάρχει μια στο δυνατόν ομαλή λειτουργία της νομισματικής πολιτικής όλη την Ευρωζώνη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες τη Ευρωζώνης και αυτό αποτελεί, ε, είναι αποτέλεσμα του ότι οι κυβερνήσεις, κάποιε από αυτές μάλλον, δεν εφάρμοσαν ε, υγιείς πολιτικές ούτε και υλοποίησαν μεταρρυθμίσεις που θα ήταν προς των πολιτών του ε, και ευρω... της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού πληθυσμού εν γέννη. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες Ευρωζώνης να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες σε εθνικό επίπεδο, ευθύνες που απορρέουν τη συμμετοχή τους στην Ευρωζώνη. Είδαμε τις διάφορες, ε, έχαμε διάφορες εμπειρίες κατά το παρελθόν, από τη δημοσιονομική εξηγήρανση που δείχνουν όμως ότι είναι σημαντικό να μειωθούν οι δημοσιονομικές ανισορροπίες και υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι για τη γιατί είναι υποφελή αυτή η δημοσιονομική εξυγίανση. Αν έχει σχεδιαστεί καλά, πρώτα απ' όλα, γιατί αν συνοδεύεται από τι κατάλληλε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, προωθεί την μακροπροθεσμή ανάπτυξη. Πρώτος λόγος. Επίσης πρέπει οι χώρες που έχουν μεγάλες ανισορροπίες στον δημοσιονομικό τομέα θα πρέπει να καταφέρουν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη. Και επίσης βοηθά να δημιουργηθούν ε, και κάποιες προστατευτικές ζώνες ε, για να αντιμετωπιστούν ε, και κάποια δίχτυα ασφαλείας για να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτα γεγονότα, απρόβλεπτες εξελίξεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αισιοδοξία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Το έχω τονίσει πολλές φορές και συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό ότι πρέπει να κάνουμε ένα ποσοτικό άλμα στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης μέσω του νομοθετικού πακέτου. Τώρα θα ήθελα να επιθυμίσω δύο σημεία. Δεν θα πρέπει να αρκεί ε, να εφαρμόσουμε ένα ισχυρότερο σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη σε τελευταία στάδια τη διαδικασία περιβολικού Θα πρέπει οι υπερβολές δημοσιονομικές να σταματήσουν νωρίτερα και να διορθωθούν νωρίτερα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος βαθμός αυτοματισμού σε πιο πρώιμο στάδιο των διαδικασιών. Δηλαδή περισσότερη ψηφοφορία με την ανεστραμμένη δική πλειοψηφία στο προληπτικό σκέλος. Και βέβαια υπάρχει και προοπτική πιο έγκαιρων κυρώσεων. Δεύτερον, θα ωφεληθούμε πάρα πολύ και από ένα εξίσου φιλόδοξο πλαίσιο μακροοικονομικών ανισορροπιών που θα λαμβάνει, θα ανοιχνεύει ε, νωρίτερα τις ανισορροπίες, θα υπάρχει αυτό το scoreboard το οποίο θα εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο και οι ανισορροπίες θα διορθώνονται έγκαιρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε εδώ στις χώρες οι οποίες τελικά δημιουργούν κίνδυνο για άλλες χώρες της Ευρωζώνης μέσω επίμονων και υπερβολικών απολύων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Να στραφώ τώρα Στι ε, σημερινέ εξελίξει ό,τι αφορά το δημόσιο χρέο. Γνωρίζετε ότι σε επίπεδο Ευρωζώνη βλέπουμε ότι η δημοσιομική εξυγένση σε πολλέ χώρε ε, εξακολουθεί και με βάση τις αρινές εκτιμήσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011 θα έχει ως αποτέλεσμα το δημόσιο έλλειμμα στην Ευρωζώνη να μειωθεί να φτάσει στο 3,5% το 2012. Αυτό είναι ενθαρρυντικό προοπτική, ιδίω αν κάνουμε μια διεθνή σύγκριση αλλά και για φέτος το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ευρωζώνης, όπως γνωρίζουμε, είναι λίγο, λιγότερο από το μισό του ελλείμματος, τον είπα και της Ιαπωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν επιλεγμένες χώρες Ευρωζώνης, οι οποίες, συγκεκριμένες ε, χώρες Ευρωζώνης, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται από μεγάλα επίπεδα χρέους και ελλείμματος. Πάντοτε η ΕΚΤ ε, καθιστά σαφές ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης ε, της ε, κατάστασης με το δημόσιο χρέος είναι μια αποφασιστική και πειθαρχημένη εφαρμογή των συμπεφωνημένων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και επίσης εφαρμογή της ατζέντα διαθροτικών μεταρρυθμίσεων για να υπάρξει μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Όσε χώρε είναι σε πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Εθνού Νομισματικού Ταμείου, ε, αυτέ οι χώρε πρέπει να εφαρμόσουν αποφασιστικά αυτά τα προγράμματα για να ε, στηθεί στα πόδια τη η οικονομία τους. Ε, αυτό ε, το αίτημα, αυτή την έκκληση την απίφθηνε άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που στην πρόσφατη συνάντησή του κάλεσε τι εθνικέ αρχέ και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ιδίω στην Ελλάδα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρά αποφασιστικά τις απαιτούμενες ε, προσπάθειες ε, ώστε η χώρα να μπει σε ένα βιώσιμο μονοπάτι. Και βέβαια γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε ε, διακομματική συνένεση και εθνική ενότητα. Έχω ξαναπεί επίσης πολλές φορές εκ μέρους και του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το χρέος συγκεκριμένα ότι είμαστε υπέρ της εθελοντικής προσέγγισης. Δεν θέλουμε πιθαναγκασμό, δεν θέλουμε καταναγκασμό. Αυτά που πρέπει να αποφύγουμε πάντως ε, είναι σίγουρα η στάση πληρωμών ή οποιαδήποτε πιστοτικά συμβάντα ή επιλεκτική πτώχευση. Ε, σίγουρα όλα αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Επίσης, ό,τι αφορά ε, τον ιδιωτικό τομέα, βλέπουμε μια κοντόθωρη αντιμετώπιση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο κινητοποιείται επίσης ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποίησεις, που είναι ένας καλός τρόπος για την κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου. Το ενθαρρύνουμε αυτό, ιδίως για την περίπτωση της Ελλάδας. όπω είπα, είναι ένα αποτελεσματικό τρόπο κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου και επιδρά θετικά και στη χρηματοδότηση τη χώρα, αλλά και σε ό,τι αφορά τι θετικέ διαθροτικέ συνέπειε για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τέλος, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, που είναι κάτι στο οποίο σκοπούν όλοι, ε, έχει ως στόχο βέβαια να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό στην αυθόρμητη χρηματοδότηση της, ε, του ιδιωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Όπως πάντα να σας θυμίσω ότι αν θέσετε μακροσκελείς και περίπλοκες ερωτήσεις θα συμβεί θα συμβούν τρία πράγματα. Ή θα σας κόψω εγώ την ε, παρέμβαση, ή δεν θα μπουν άλλοι στον κατάλογο για να, βάλουν την, για να θέσουν ερώτηση, ή δεν θα πάρετε απάντηση από τον πρόεδρο. Οπότε γενικώ προσπαθήστε να είσαστε έτσι συνοπτικοί για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε όλοι από την παρουσία του πρόεδρου. Και για να μην έτσι με εξαγριώσετε και εμένα. Πρώτη ερώτηση από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν θέσω το ερώτημά μου, θα ήθελα να σας, να σας συγχαρώ για την απονομή του ε, βραβείου Καρλ. Είναι νομίζω εξαιρετικό, είναι μεγάλη τιμή αυτή για έναν μεγάλο Ευρωπαίο. Τώρα, πάω στο ερώτημά μου. Για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Πώς αξιολογείτε εσείς την πρόταση Τη γαλλική κυβέρνηση για τη συμμετοχή των ιδιωτικών, του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ δύο πράγματα με ενδιαφέρουν κυρίω. Ένα, έχετε ήδη κάποιο feedback, κάποιες έτσι απαντήσεις από τους οίκους αξιολόγησης για τις τεχνικές ε, λεπτομέρειες, γιατί αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την υπόθεση την, ε, της οικονομικής ε, Ήδη ο Σόιμπλε είπε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την επιρροή που έχουν αυτοί οι οίκοι αξιολόγηση. Και αν δούμε ότι ας πούμε οι συνεργάτες της ε, ε, Fitch γράφουν στα, στον, στις New York Times και ότι συνέχεια υπάρχουν αλλαγές στις ε, προθεσμίες. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε εις βάθος. Ένα δεύτερο πράγμα που με απασχολεί Μάλλον αντιτίθεται λίγο στην πρόταση αυτή το δεύτερο, δηλαδή η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για τον ηθικό κίνδυνο. Ε, σε αυτή την σε αυτή την προσπάθεια θα μπουν όντω αρκετοί ιδιώτες επενδυτές και επίσης μήπως υπάρξει περίπτωση να δημιουργηθούν ε, προηγούμενα για μελλοντικέ υπερχρεώσεις από κάποια κράτη-μέλη. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας ε, λόγια. Με συγκινείτε. Για το πρώτο σας ερώτημα, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το θέμα αυτό των συζητήσεων της ε, εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα μεταξύ των κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα, είναι ευθύνη των κυβερνήσεων. Εμείς βεβαίως παρακολουθούμε την κατάσταση πώς εξελίσσεται. Όπως είπα, έχουμε δώσει και τη δική μας ε, συμβουλή. Να μην είναι δηλαδή υποχρεωτικές αυτή, να μην είναι υποχρεωτική η συμμετοχή, να αποφύγουμε την χρεοκοπία, να αποφύγουμε τα πιστωτικά, ε, ε τα τις πιστοτικές περιπτώσεις αυτές, αλλά ε, αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων, το οποίο θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε προς το παρόν, επαγρυπνούμε, παρακολουθούμε το τι γίνεται, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω μια πολύ συγκεκριμένη εκτίμηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ξέρω βεβαίως ότι ακόμη υπάρχουν θέματα ανοιχτά για την φύση, ας πούμε, του, της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Τώρα, ένα σημαντικό ακόμη θέμα είναι να αναφερόμαστε στην, 28, στην ε, συμφωνία της 28 Νοεμβρίου μεταξύ των μελών του Eurogroup που δημοσιοποίησαν το δόγμα τους σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Το κείμενο αυτό που είναι πολύ σημαντικό και έχει δημοσιευθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ως ε, παράρτημα στη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μετά τη συμφωνία αυτή της 28 Νοεμβρίου λέει σαφέστατα πως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπως ας πούμε το δόγμα του IMF, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδέα είναι ότι με τις απαραίτητες προσαρμογές θα πάμε πίσω σε εθελοντική χρηματοδότηση της αγοράς. Αυθόρμητη ε, χρηματοδότηση της αγοράς με κάποια προσαρμογή βεβαίω. Όπου δηλαδή δεν υπήρχε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με την ε, έννοια της αναδιάρθρωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια θα δείτε ότι η κρίση της ε, Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας είναι ότι αυτό μπορεί να μην γίνεται, να μην είναι εφικτό. Αλλά εγώ σας παραπέμπω στο διεθνές δόγμα που υιοθέτησε το Eurogroup στο τέλος του Νοέμβρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ο Εντουάρτ για τους σοσιαλιστές. Προσωπικούς χαιρετισμούς, κύριε Τρίσε, και από το συντονιστή της ομάδας με τον κύριο Μπουνά. Τώρα, αν δούμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κρίση. Χρησιμοποίησε ε, ουσιαστικά αυτορμητισμό Δεν είχαμε σχέδιο και ασκήθηκε κριτική γιατί κάθε φορά οι απαντήσει ε, και διορθώσεις ε, δίνονταν πολύ καθυστερημένα. Τώρα αν ε, ξεκινούσαμε από την αρχή, άλλωστε την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και αυτό υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Τι θα λέγατε, να περιλάβουμε το εξή, όχι σε σχέση με την πρόληψη των κρίσεων. Έχουμε συμφωνήσει επ' αυτού, αλλά για τους πιο δύσκολα τμήματα της πρόληψης ε, των κρίσεων, εμείς θεωρούμε ότι στην ομάδα μας ε, δεν υπάρχουν ιδέες για ε, την ανάπτυξη της οικονομίας. Ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες, παραδείγματος χάρη, συνοδεύτηκε από χαμηλά επιτόκια και άλλα συνοδευτικά μέτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβα ότι επικεντρώνετε την ερώτησή σας ε, στη διαχείριση της ε, κρίσης και όχι στην πρόληψη της κρίσης, αλλά και η πρόληψη της κρίσης είναι ε, ουσιαστική και αν μπορούμε κάτι να συμπεράνουμε από τα σημερινά γεγονότα είναι ότι πρέπει να επιβάλλουμε μέτρα, πρέπει να βελτιώσουμε την πρόληψη της ε, κρίσης από το Συμβούλιο το 2004 και το 2005 μεγάλες χώρες Όλες ε, οι μεγάλες χώρες ήταν υπέρ της ε, αποδυνάμωσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης Δηλαδή ήθελαν να καταργήσουν τα κυρία στοιχεία του συμφώνου και υποστηρίχθηκαν πάνω κάτω από ε, αρκετούς οικονομολόγους. Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρό. Και βλέπουμε τώρα ε, ποια είναι τα αποτελέσματα. Από το 2005 η ΕΚΤ έλεγε ότι πρέπει πολύ προσεκτικά να ε, παρακολουθήσουμε τις ανισορροπίες ε, στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα και σε επίπεδο 27 κρατών μελών ε, αλλά και την ανταγωνιστικότητα. Τώρα αυτό έχει γίνει αποδεκτό βάσει της κρίσης, λόγω της κρίσης. Όμως ξέρουμε ότι έχουμε δύο δυσκολίες σήμερα. Έχουμε τη δημοσιονομική πολιτική και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του, της κρίσης, ε, ξέρετε ότι ο EFSF και το ESM ε, θέλουμε να είναι όσο δυνατόν πιο ευέλικτα και καλούμε η προσαρμογή να είναι το δυνατόν πιο αξιόπιστη και πιο σταθερή. Να το δυνατόν πιο πάγια, γιατί θέλουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι μια έννοια, ε, ξέρετε, πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών, των επενδυτών, των αποταμιευτών, του οίκου και φυσικά όλα αυτά βασίζονται στις αποφάσεις που λαμβάνει κανείς και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν να αυξηθεί το δυναμικό της ανάπτυξης και για τα μέσα που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης καλούμε να έχουμε μέγιστο βαθμό ευελιξίας. Εμείς έτσι ε, σκεφτόμαστε, δίνουμε αυτές τις συμβουλές, αλλά φυσικά ε, τα κατάλληλα όργανα και οι κατάλληλοι θεσμοί πρέπει να λάβουν αυτές τις αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τους ελεύθερου, Σιλβί. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καταρχήν ένα σχόλιο. Εμένα την τελευταία εβδομάδα με εξέπληξαν οι ταυτόχρονε διαπραγματεύσει για την οικονομική διακυβέρνηση και τη διαδικασία διορισμού του διαδόχου σα. Έχουμε την εντύπωση για τα κρατημέλη ότι υπάρχουν κάποιοι άγραφοι κανόνε, οι οποίοι μετράνε πάρα πολύ και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και ίσω να περιορίσουμε για κάπω την ανεξαρτησία τη ΕΚΤ και υπάρχουν και κάποιοι κανόνε που ε, δεν ε, μπορούμε να μην τους σεβαστούμε. Ε, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ε, θεωρώ ότι ε, όταν προσπαθούμε εδώ με εθνικές ε, υπεράσπιση εθνικού συμφερόντος να παραβιάζουμε το ευρωπαϊκό συμφέρον είναι πραγματική επίθεση. Τώρα, πέραν αυτών για τους γραπτούς κανόνες, ε, γιατί, κοιτάξτε, αυτούς ε, θέλουν να σέβονται ε, οι άνθρωποι τους γραπτούς κανόνες. Σας ευχαριστώ που είπατε στην παρουσίασή σας ότι χρειάζεται οπωσδήποτε περόληψη και μεγαλύτερη αυτοματισμοί. Ακούσατε κ. υποκυριολόγηση και την περασμένη εβδομάδα. Πιστεύετε ότι αν δεν έχουμε τέτοιου είδου στοιχεία ε, θα έπρεπε να μείνουμε με το σύμφωνο όπως είναι μεταξύ του Quantum Leap και του Leap Service, λέω μιλήτρια στα αγγλικά, εγώ προτιμώ το Quantum Leap. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξαρτησία της ΕΚΤ, ε, ξέρετε ότι εμείς ε, έχουμε πολύ ξεκάθαρα καθορίσει την ανεξαρτησία μας. Όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των μεγάλων χωρών μας ζήτησαν να μειώσουμε τα επιτόκια το 2004, είπαμε όχι. Θα θυμάστε ε, ότι εμείς είχαμε 2%, όταν είπα είχαν 1% και εμείς είπαμε όχι. Και είχαμε αίτημα που προερχόταν από τρεις μεγάλες χώρες από αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Εμείς αυξήσαμε τα επιτόκια στα τέλη του έτου 2005, το Δεκέμβριο, ενώ 10 κυβερνήσει στις 12 τότε διαμαρτύρονταν δημοσίω και έντονα. Και θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα της αποφασιστικότητάς μας, φυσικά συμπεριλαμβάνεις και τις διαμάχες που είχαμε το 2004 και το 2005, όπως και η Κομισιόν με τις κυβερνήσεις που ήθελαν να διαλύσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ε, είπαμε όχι στο Συμβούλιο των Κυβερνώντων ότι είχαμε grave concerns, πολύ μεγάλες ανησυχίες σε σχέση με τόσο συνέβαιναν και ε, ήταν ε, ακόμη πιο ε, σοβαρό και δεν επρόκειτο για το γράμμα του νόμου αλλά για την ουσία. Και εσείς αναφερθήκατε σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τις σημερινές διαπραγματεύσεις, δεν έχω συμβουλές να σας δώσω. Έχει τοποθετηθεί σχετικά το Κοινοβούλιο. Βρίσκεται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης στον τριμερή διάλογο. Είμαι επιπισμένος ότι το Κοινοβούλιο ακολουθεί ένα προσανατολισμό που είναι ορθός προς το συμφέρον της Ευρώπης, νομίζω ότι η ιστορία θα μας, θα μας κρίνει όλους και μάλιστα αυστηρά. Θα κριθούν και οι θεσμοί που ήταν αδύναμοι στο να συνειδητοποιήσουν τα διδάγματα της κρίσης. Η παγκόσμια κρίση μας αποκαλύπτει κάποιες αδυναμίες, είναι αλήθεια το να μην τις ε, διορθώνουμε τόσο γρήγορα όσο χρειάζεται και πλήρως είναι βαριά ευθύνη. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και εντάσεις ε, μεταξύ εθνικών ανησυχιών και ευρωπαϊκών ανησυχιών. Εμείς είμαστε ένας ευρωπαϊκός θεσμός και εσείς είστε ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ένα ευρωπαϊκό όργανο. Εμείς ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε κάπου να συναντηθούμε σε τέτοια θέματα και έχουμε πει επανειλημμένω ότι στο πλαίσιο της σημερινής συνθήκης, γιατί δεν ε, πρόκειται να αλλάξουμε τη συνθήκη αμέσως, ακόμη και αν αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάμε στο δυνατόν λοιπόν πιο μακριά στην ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τώρα, αν έλεγα ότι ε, η σημερινή κατάσταση δεν είναι καλύτερη από το προηγούμενο Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη, δεν υπερέβαλα. Έχουμε προσθέσει και τους δείκτες για την ανταγωνιστικότητα και για την αντιμετώπιση των ισορροπιών. Και αυτός είναι σημαντικός δεύτερος πυλώνας. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι, αλλά αν ε, συγκρίνουμε αυτή την πρόοδο με το ότι δεν φτάσαμε μέχρι το τέρμα, είναι πολύ σοβαρό κατά την άποψή μας και ελπίζω διακαώς ότι θα καταλήξετε αποφασιστικά σε μια καλύτερη λύση από τη λύση που μας προτείνετε σήμερα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Και okay, παρακαλώ εκ μέρους της CCR. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο ηγηθήκατε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εν μέσω μιας σημαντικής οικονομικής κρίσης, ε, ύφεση ε, και μεγάλου προβλήματος με την φερεγγιότητα και την ρευστότητα. Με τις όλες προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία νομίζω ότι καλά ε, τα έχουμε καταφέρει, νομίζω έχουμε αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και πρέπει να σας ε, απονείμουμε τα εύσημα γι' αυτό κύριε Τρισέ. Τώρα, υπάρχουν πρόσφατες εκθέσεις που λένε ότι η Κίνα προσπαθεί να επενδύσει περισσότερο ε, σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ και όχι τόσο ε, στο δολάριο πλέον. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, στην καμπύλη απόδοσης ε, του δολάριου στις ΗΠΑ μία πτωτική τάση και βλέπουμε ότι μειώνονται οι αποδόσεις κατά των θεμελιωδών οικονομικών. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάτι αντίστοιχο στις ευρωπαϊκές πιστώσεις. Υπάρχουν κάποια αρνητικά τα οποία θα αντιστάθμιζαν τα θετικά στοιχεία της επένδυσης αυτής. Η απάντηση είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Uh, uh, Πραγματικά τα πάντα είναι ανοιχτά αυτή την εποχή και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι επενδυτές, αποταμιευτές αναλύουν και κρίνουν επιμονή μου βάσεως ε, ποια είναι η καλύτερη επένδυση στην οποία θα μπορούσαν να προβούν. Όπω γνωρίζετε και εμείς οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ποτέ δεν ξεκινήσαμε κάποιο είδου παγκόσμια εκστρατεία υπέρ της επένδυσης, ε, υπέρ του ευρώ τους επενδυτές. Θεωρούσαμε πάντοτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίζεται, θα έλεγα, αποκεντρωμένα. Δηλαδή, από κάθε αποταμιευτή, από κάθε επενδυτή. Βέβαια, τούτου λεχθέντος εκτιμώ όλο ιδιαίτερω αυτό που είπατε. Δηλαδή ότι πράγματι αποκαταστήσαμε την εμπιστοσύνη και αυτό αντικαθρεπτίζεται ξεκάθαρα στο ευρώ. Και αυτό δεν με εκπλήσει, ξέρετε, διότι το παράδοξο της Ευρωζώνης ή του ευρώ είναι ότι ναι, μην υπάρχουν προβλήματα, έχουμε προβλήματα, δεν θα πρέπει να είμαστε αυτάρισκοι σε καμία περίπτωση απέναντι στα προβλήματα αυτά διακυβέρνηση ή κάποια προβλήματα μεμονωμένων χωρών. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν δείτε την προοπτική συνολικά τη Ευρωζώνη, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά. Έχουμε ίσως και τρέχουμενου ε, τρέχουμενους για την Ευρωζώνη συνολικά. Έχουμε μεν αυτό το έλλειμμα των δημόσιων οικονομικών, αλλά όπω είπα είναι το μισό του ελλείμματος άλλων προηγμένων παγκόσμιων οικονομιών, όπως είναι είπα η Ιαπωνία, έχουμε ανάπτυξη που έχει επιβεβαιωθεί μάλιστα και επιβεβαιώνεται κάθε τρίμηνο και μάλιστα η αναθεώρηση είναι πάντοτε επιτάνω σε σχέση με τα προβλεπόμενα. Και στην εισαγωγική μου παρατήρηση μίλησα για τις τελευταίες μας προοπτικές που τελικά έβαλαν πιο ψηλά, ε, κατά 0,3% το ποσοστό σε ό,τι αφορά τις ε, νέες μας προοπτικές. Και βέβαια και το νόμισμα έχει διατηρήσει ε, με εκπληκτικό τρόπο, θα έλεγα, την αξία του τα τελευταία 12 ε, χρόνια, με τον πληθωρισμό να κινείται γύρω στο 2% τελευταία. Αυτό ισχύει, επαναλαμβάνω, για όλη την Ευρωζώνη, ένας υπολογισμό που αφορά την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Και ξέρετε ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι το καλύτερο από οποιοδήποτε κράτος μέλος Ευρωζώνης ατομικά για οποιαδήποτε δωδεκαετία κατά τελευταία 50 χρόνια. Επομένως είναι ε, πάρα πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα αυτά. Και βέβαια συμβαδίζουν με το βασικό στόχο μας και την εντολή που έχουμε βασικά. Δεν θέλω να ε, κάνω συγκεκριμένα σχόλια. Ε, τώρα σε αφορά την Κίνα συγκεκριμένα, βέβαια μπορώ να πω ότι και αυτοί κοιτούν πώς θα βελτιστοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις τους και τις οικονομίες τους τις αποταμιεύσεις τους. Την ίδια στάση έχουμε απέναντι στους Κινέζους ε, με αυτή που έχουμε και απέναντι σε όποιον άλλο πιθανό επενδυτή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, ο Φίλιπ. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε για ρευστότητα, για αφαιρεγκαιότητα εξακολουθείτε να επιμένετε ότι το ελληνικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα ρευστότητα ε, και όχι αφαιρεγκαιότητα. Ο συνάδελφό σα, Μέρβιν Κίνγκ, λέει ακριβώ το αντίστροφο. Δεν ξέρω, τα λέτε ποτέ μεταξύ σα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλο πάντων, αν το πρόβλημα, το ελληνικό δεν είναι πρόβλημα αφαιρεγκαιότητα, υπάρχουν προβλήματα αφαιρεγκαιότητα. Ή με άλλα λόγια, τι θα σας οδηγούσε να κρίνετε αφαιρέγγιο ένα κράτος μέλος και αν η Ελλάδα δεν Εμπίψα αυτή την περίπτωση, πώς εξηγείται τα επιτόκια που πρέπει σήμερα, μάλλον τους στόχου που πρέπει σήμερα να καταβάλει, αν ε, θέλει να επιστρέψει στι ε, αγορές. Και κάτι δεν κολλάει εδώ. Ο ιδιωτικό τομέα λαμβάνει ε, κάποια επιτόκια, περιλαμβάνουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου για ένα κίνδυνο που δεν υπάρχει. Τελικά μιλάμε για μεταφορά του πλούτου από το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες στους ιδιώτες πιστωτές. Επομένως βλέπω ότι δεν ε, ε, υπάρχει συμβατότητα σε όλα αυτά που λέτε. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αν έχει την καλοσύνη αυτό. Je vous dirai, να σας πω καταρχήν ότι η επιτυχία μιας προσαρμογής είναι η επιστροφή στην εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτό θεωρώ επιτυχία σε παγκοσμίο επίπεδο. Είναι στιγμή που οπότε οι αγορές ε, αυθόρματα, δηλαδή οι επενδυτές αυθόρμητα επανέρχονται γιατί έχουν εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη δεν ενθαρρύνεται τόσο αν ε, τελικά μας ενθαρρύνεται μόνιμα να κάνουμε μία συζήτηση για το αν ε, θα πρέπει να έχουμε ένα πρόβλημα φερικιότητας ή ρευστότητας. Αυτό ήδη αποφασίστηκε από τη διεθνή κοινότητα τη στιγμή που θετήθηκε για πρώτη φορά το σχέδιο για την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν για μια ακόμη φορά το σίγουρο είναι, το βέβαιο είναι ότι αν υπάρχει μία αέναη συζήτηση τότε δεν κάνουμε όσο είναι απαραίτητα για την επιτυχία και όλοι έχουμε συμφέρον για την επιτυχία και η Ελλάδα και οι γείτονες της Ελλάδας, ε, όχι μόνο οι χώρες της Ευρωζώνης ε, και ούτε μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν σας ενθαρρύνω να λάβετε αυτή τη συζήτηση πάρα πολύ σοβαρά και εγώ θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με λιγότερο θεαματικό τρόπο βέβαια από τη σήμερα και αφού θα έχει ληφθεί ε, μια υπόφαση θα ήθελα και να στέκει. Τώρα, η κατάσταση με τον ιδιωτικό του κομμέα είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι πιστεύετε. Αν τα επιτόκια βρίσκονται στο επίπεδο που γνωρίζετε, αυτό συμβαίνει επίσης γιατί ορισμένοι δεσμεύτηκαν, ανέλαβαν ε, κάποιες ε, συναλλαγές ε, που κινούνται είτε από το φόβο, δηλαδή φοβούνται μήπως χάσουν χρήματα ή έχουμε την καθαρή κερδοσκοπία. Δηλαδή να κάποιοι θέλουν να κερδίσουν χρήματα γιατί μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενη χοροκοπια Έτσι λοιπόν να θεωρήσουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο πολύπλοκος σήμερα από ότι 20 χρόνια πριν έχετε ουσιαστικά ε, κάποιους ε, ε, ομιλίες μακροσκελής και το αντίθετο τώρα. Ε, ίσως ε, θα πρέπει ε, Τώρα εδώ να μην ωφελήσουμε τους κερδοσκόπους γιατί αν το κάνουμε αυτό θα βρεθούμε σε μια παράδοξη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, εμείς ε, ενθαρρύνουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποφασιστικοί. Η προσαρμογή της χώρας είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει και το λέω ξεκάθαρα. Από αυτή τη σκοπιά είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε σε όλες τις χώρες που έχουν ένα πρόγραμμα, αξιόπιστο πρόγραμμα προσαρμογής, ικανό να πείσει το σύνολο των παρατηρητών και φυσικά των ενδεχόμενων επενδυτών και επίσης ε, να υποστηρίζεται ευρέως από την ίδια τη χώρα. Αναφέρθηκα επίσης ότι χρειάζεται και μια ευρεία ένωση όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που διακυβεύεται το σύνολο της χώρας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τα πράγματα με αποφασιστικό τρόπο και με όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρο τρόπο. Τώρα, στην περίπτωση της Ελλάδας, η πρώτη προϋπόθεση είναι το ίδιο το πρόγραμμα, το ίδιο το σχέδιο. Φυσικά συζητούμε το ότι λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Και η δεύτερη προϋπόθεση που είναι σημαντική για την ελληνική περίπτωση είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Είπα και κάτι στην εισαγωγική μου παρέμβαση για τις ιδιωτικοποίησεις η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες έχει αυτό το πλεονέκτημα, κατέχει αυτό το πλεονέκτημα. και έχει την ικανότητα να ιδιωτικοποιήσει, να ενεργοποιήσει ιδιωτικά κονδύλια βάσει σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων γιατί έχουμε σήμερα 50 δισεκατομμύρια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, δηλαδή περίπου 20% του ΑΕΠ. Είναι μεγάλο το ποσό. Αλλά, συμπερασματικά, είναι προς το συμφέρον του ελληνικού έθνους και του ελληνικού λαού να γίνει κάτι τέτοιο για να δημιουργηθούν θέσεις ε, εργασίας, μεσοπρόθεσμα, ε, και φυσικά αυτό ενδιαφέρει και όλη την διεθνή κοινότητα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Η εμπιστοσύνη να μπορέσει να επανέλθει το συντομότερο δυνατό και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι ο καθένας ε, από εμά έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει σε αυτή την εμπιστοσύνη που πρέπει να ανακτηθεί. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, της ΓΟΥ, κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή ενημέρωση που μας κάνετε. Άλλωστε, εκτιμώ πολύ ότι μας δίνετε και γραπτά την εισήγησή σας, με συνέπεια να μπορεί κανείς να επανέλθει, αν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν θα σας ρωτήσω για την Ελλάδα, γιατί μοιάζει λίγο κουραστικό. Ήδη δώσατε κάποιες απαντήσεις. Αναφερθήκατε για κάποιους δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη και το δημόσιο έλλειμμα. Έχουμε όμως τρεις χώρες. Την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία που είναι στο μηχανισμό στήριξης και εφαρμόζουν προγράμματα λιτότητας. Για την Ελλάδα τα ξέρω. Δεν το εφαρμόζει, δεν έχει εθνική συνένεση, μπορεί να κάνει αυτό κτλ. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν είναι σωστά αυτά που διαβάζω στον τύπο, σχετικά με τα αποτελέσματα στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Και τι θέλω να σας πω. Τα στοιχεία λένε πως οι χώρες βυθίζονται και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία σε ύφεση, με συνέπεια να μεγαλώνουν τα ελλείμματα και να χρειαστούν νέο δανεισμό καθώς το χρέος θα αυξηθεί. Η ερώτηση κύριε Τρισά είναι απλή. Στην Ελλάδα φταίει τόνα. Στην Ιρλανδία δεν ξέρω τι φταίει. Στην Πορτογαλία δεν ξέρω τι φταίει. Μήπως δώσαμε λάθος φάρμακο στους ασθενείς. Και μια πιο απλή ερώτηση. Στην περίπτωση που έχουμε νέο δανεισμό όπως συζητείτε για την Ελλάδα, με την εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών. Από τα όσα διαβάζω, εκεί θα υπάρχει και μια επιδότηση επιτοκίου, δηλαδή θα δοθεί κάποιο κίνητρο στους ιδιώτες για να ανταλλάξουν τα ομόλογα. Θα ακολουθηθεί μια τέτοια πολιτική. Θα κάνετε κι εσείς μια τέτοια πολιτική επιδότηση του επιτοκίου στις τράπεζες για να συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική ανακύκλωση των ομολόγων. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Κάποια σχόλια για το ερώτημά σας, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε λιτότητα είναι ουσιαστικά η διόρθωση κάποιων εξελίξεων πολλών στο παρελθόν που δεν ήταν λογικές και θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Δεν θέλω τώρα να σας ζαλίσω με πολλά νούμερα, αλλά ο, ο μέσος όρος ανάπτυξης του κόστους, αύξηση του κόστου στις τρεις χώρες που μας αναφέρατε ήταν πάρα πολύ υψηλότερος από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης. Ας πούμε, μισθή στο δημόσιο τομέα με το ίδιο νόμισμα, το ευρώ ίδιο κόστος διεθνώς, γιατί είναι το ίδιο νόμισμα. Η ίδια ε, διεθνής αγοραστική δύναμη, γιατί είναι το ίδιο νόμισμα. Με το ευρώ μπορείς να αγοράσεις το ίδιο πράγμα παντού στον κόσμο. Είτε είσαι σε αυτές τις τρεις χώρες που αναφέρατε, είτε είσαι σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Μισθή λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση το πρώτο, τα πρώτα τρία χρόνια από ό,τι θυμάμαι ήταν περίπου 38%. Σε κάποιες χώρες ήταν πολύ μεγαλύτερη. Σε δύο χώρες έφτανε πάνω από το 100%. Οπότε δεν ήταν λογικό. Και εμείς έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια να λέμε ότι δεν είναι λογικό αυτό που γίνεται, δεν είναι λογικό, δεν είναι λογικό. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η διόρθωση όχι κάτι που έρχεται από κάποια αφηρημένη έννοια και επιβάλλεται για αφηρημένους λόγους. Όχι, διορθώνουμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Και αυτές οι διορθώσεις είναι απαραίτητες εάν θέλουμε να επανέλθουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης και σε δημιουργία θέσεων εργασίας. Μία χώρα, πρέπει να πω, δεν θέλω να συγχαρώ βεβαίω κάποια χώρα ιδιαίτερα. εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλη την Ευρωζώνη και καταφέραμε να έχουμε ένα 2% για το σύνολο της Ευρωζώνης. Αυτό μας ζητείτε να κάνουμε και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Πρέπει να έχετε βέβαια υπόψη σας ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την Ευρωζώνη στο σύνολό της. Εγώ είμαι στη θέση του Μπερνάγκη ας πούμε δεν μπορώ να... Ο Μπερνάγκη όπως δεν μπορεί να ασχοληθεί με το αν η Αλάσκα ή η Νεβάδα έχει ειδικό συγκεκριμένο πρόβλημα, με το ίδιο πράγμα, δεν... με το επιμέρους πρόβλημα δεν ασχολούμαστε κι εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις κυβερνήσεις που βρίσκονται στην Ευρωζώνη. Οι υπόλοιπε αρμοδιότητε μα είναι η εποπτεία τη Ευρωζώνη, η εποπτεία, ας πούμε, η παρακολούθηση των δράσεων τη Κομισιόν, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για οι μεμονωμένε συμπεριφορέ των χωρών. Εμεί δίνουμε τη συμβουλή μα και σα το λέω ξεκάθαρα. Αυτή είναι η δική μα ευθύνη. Αυτή λοιπόν η χώρα που ήταν πάρα πολύ προσεκτική που φρόντισε να μην χάσει ανταγωνιστικότητα ή τέλος πάντων που ήθελε να ξαναέχει ανταγωνιστικότητα έδωσε πάρα πολύ προσοχή στο κόστος της μονάδας. Γιατί όλες οι, όλοι γνωρίζουμε ποιες, ποιες είναι, ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό που θέλουμε σήμερα είναι η ανάπτυξη, είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και είναι και η αντίσταση. Έχουμε, βρισκόμαστε στην χειρότερη κατάσταση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε είναι σαφές ότι το να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται τα πράγματα καλά είναι ο δρόμος για να φτάσει στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, ε, πρόκειται να, γίνουνε να ξαναγίνουν τα, τα stress των τραπεζών. Όταν ε, έγινε το ίδιο πράγμα το προηγούμενο χρόνο, βρέθηκαν 7 από 99 που απέτυχαν, από 91 τράπεζε μάλλον που απέτυχαν το τεστ. Οι υπόλοιπε που πέρασαν έπρεπε να επανακρατικοποιηθούν. Αυτό υπονομεύει την ίδια την ουσία των τεστ. Τα τεστ τα καινούργια, από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνουν υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Αλλά τώρα είναι αρκετά ρεαλιστικό να δούμε αν υπάρχουν και ε, τραπέζες που δεν έχουν κρατικοποιηθεί. Και Επίσης, το θέμα της ελληνικής χρεοκοπίας και της Ιρλανδικής και της ε, ε, Πορτογαλικής θα πρέπει να το δούμε. Η... Ποια είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στην ευρωπαϊκή κρίση. Έχετε υπολογίσει τι θα σημαίνει μια, ευρωπαϊκή, μια ελληνική συγγνώμη, χρεοκοπία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πόσο, πόσο, τι, τι μέγεθο απώλεια μπορεί να απορροφήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να τους, πριν γυρίσετε στα κράτη-μέλη και ζητήσετε και άλλο κεφάλαιο. Και επίση, είσαστε πολύ συνετό τραπεζίτη. Τι θα λέγατε σε, ένα, σε έναν πελάτη που θα, που θα ερχόταν να σα πει ότι δεν μπορεί να πληρώσει του λογαριασμού του τον επόμενο μήνα, αν σα έλεγε ότι έχει χρεοκοπήσει τελείω και ότι, δεν, ε, ότι έχουν μείνει τα, οι δύο τα δύο τελευταία του ευρώ και τα τελευταία, τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να πληρώσει. Τι θα του λέγατε, θα του έλεγατε να πάει να δανειστεί κι άλλο και να αυξήσει κι άλλο, στο, κι άλλο το χρέος του. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, είπατε, είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών υπεύθυνη για αυτά τα τεστ αντοχής, ε, για αυτά τα stress test και έχουν γίνει με τον ε, καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα δούμε πότε θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα των τεστ, των δοκιμών αυτών, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν θέλω εγώ να προτρέχω από τη δουλειά που έγινε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τροπεζών και από όλους ε, τους εθνικούς επόπτες, γιατί ξέρετε ότι πρόκειται για ένα έργο που γίνεται και με την συμμετοχή των εθνικών εποπτικών αρχών. Δεύτερο σχόλιο. το οποίο πάντα και στη δεύτερη ερώτησή σα. δεν είμαστε <laughs> στι Ηνωμένε Πολιτείε. δεν είμαστε Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε έχουμε ε, μία νέα Υπουργείο Οικονομικών, ε, μία ομοσπονδιακή κυβέρνηση και μία νέα υπογραφή. Έχουμε 27 κυβερνήσεις, 27 υπογραφές ε, και 27 κράτη που πληρώνουν φόρους. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα Θέλουμε να έχουμε και έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, θέλουμε να έχουμε μια αγορά για τους 27 και όπως ξέρετε αυτά τα stress test γίνονται σε επίπεδο 27 κρατών μελών. Το γεγονό είναι ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός αντιστοιχίας ε, μεταξύ της, ε, επιτροπή, της, της υπογραφής ε, των ε, τραπεζών και του προπολογισμού σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Και αν υπάρχουν και των κυβερνήσεων και αν υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο κράτους, τότε υπάρχουν και προβλήματα σε επίπεδο τραπεζών. Γιατί ξέρετε, αν υπάρχουν προβλήματα δημοσιονομικά στο κράτος, τότε ε, υπάρχει πρόβλημα στα μάτια των επενδυτών για την ενδυνάμει σταθερότητα των τραπεζών. Γιατί μειώνεται η αξιοπιστία ή αρχίζουν τα ερωτηματικά σχετικά ε, με τη σταθερότητα των δημοσιονομικών του κράτους. Και έτσι λοιπόν πάντοτε πρέπει να θυμόμαστε σε ποιο συσχετισμό ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις οι δημοσιονομικές ε, για την Ευρώπη. Είμαστε μία ενιαία αγορά με ένα ενιαίο νόμισμα, ενώνουμε 300-350 εκατομμύρια άτομα μέσα στα 500 εκατομμύρια, όμως ε, παρόλα αυτά έχουμε ένα σύνολο και κυβερνήσεων και κοινοβουλίων. Θα έλεγα λοιπόν μόνο ως ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμείς ε, ε, κόβουμε νόμισμα για 17 χώρες. Και για τις 17 χώρες, όχι μόνο για ένα τμήμα των 17. Αυτά τα καθήκοντα μας εναποθέτει η συνθήκη και έχουμε και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δίνουμε απαντήσεις, ε, έχουμε ένα πλαίσιο για τις ασφάλειες, είναι απόλυτα δημόσιο αυτό. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αυτό είναι βελτιστοποιημένο. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε τα πρότυπα μέτρα, δηλαδή τα μέτρα για το επιτόκια που λαμβάνουμε για να έχουμε σταθερότητα των τιμών και τα μη πρότυπα μέτρα, τα οποία λαμβάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι αντιμετωπίζουμε τη μη ομαλή λειτουργία ορισμένων αγορών. Αυτά πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε. Φυσικά, Ζούμε τώρα τα αποτελέσματα της χειρότερης παγκόσμιας κρίσης μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπορούσε να είναι η χειρότερη ε, κρίση και από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι πάρα πολύ σοβαρή λοιπόν. Έτσι λοιπόν θα υπενθυμίσω ότι είπαμε την ε, περασμένη φορά ότι είμαστε σε κατάσταση ε, έντονης εποπτείας ισχυρή εποπτείας και είπαμε ότι θα διατηρήσουμε ε, το σταθερό επιτόκιο για ε, το τρίτο τετράμινο του έτους και θα δείξουμε ότι έχουμε εφαρμόσει την αρχή του διαχωρισμού, δηλαδή μεταξύ των πρότυπων μέτρων και των μη πρότυπων μέτρων και να σας πω ότι εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε σταθερότητα των τιμών στο χρόνο. Συνεχίζουμε να το πράττουμε αυτό. Αυτό είναι κάτι που για μας είναι απολύτως θεμελιώδες. Είναι η συνθήκη, αυτό που μας καλούν οι λαοί να πράξουμε και είναι ουσιαστικό για τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη της στην Ευρωζώνη στο σύνολό της, προκειμένου να διατηρήσουμε την ευμερία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ και τώρα για το ΕΛΚ. Αντιπρόεδρος Χωσέ Μανουέλ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που θα πούμε στο επανειδήν και εγώ θέλω να θέσω μια πολύ γενική ερώτηση σε εσά που είστε και φιλοευρωπαίο και ανεξάρτητο αμερόληπτο. Ξέρουμε ότι η νομισματική ένωση δεν ήταν βέλτιστη ε, νομισματική βελτιστώς νομισματική περιοχή. Έχουμε φυσικά το σύμφωνο σταθερότητας και ο συντονισμός των διάφορων πολιτικών θα επέτρεπαν ε, να εξελιχθούν οι μεγαλύτερες διαφορές ε, μεταξύ των διάφορων κρατών μελών, όμως αυτό δεν έγινε ούτε στους καλύτερους ούτε στους χειρότερους καιρούς ε, και δεν ε, ε, έχουμε σεβαστεί οι τρεις βασικές αρχές του no bailout, του no default και θα μπορούσαμε να αποτύχουμε και στο no exit. Ε, δηλαδή, ε, εσείς αναφερθήκατε και σε μια πιθανή τροποποίηση της συνθήκης. Ε, ο κύριος Δράγκη αναφέρει τη δυνατότητα των ευρωομολόγων, δεν το αποκλεί. Και ο κύριος Τρισέ είπε ότι δεν είναι αδύνατο μέσα στην θεσμική αρχιτεκτονική. Δεν είναι δυνατό, αλλά αν η ιδέα είναι καλή θα έπρεπε να αλλάξουμε αυτή την ε, θεσμική αρχιτεκτονική. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε και να ελπίζω να έχουμε και την ε, δική σας εμπειρία τα επόμενα χρόνια και φυσικά για τους επόμενους μήνες θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για, και να μας βοηθήσετε στον δρόμο στον οποίο θα ακολουθήσουμε με την εμπειρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην πολυμορφία της κατάστασης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Και πράγματι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Κάποια στιγμή θα συγκλίνουμε, αλλά δεν έχουμε ακόμη επαρκώς συγκλίνει. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς ε, στην έρευνα που κάνουμε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή την πολυμορφία σε μια προηγμένη οικονομία. Μπορούμε να συγκρίνουμε τη ΣΥΠΑ με την Ευρωζώνη για μια ακόμη φορά. Αυτό το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει είναι ότι στη ΣΥΠΑ βλέπουμε ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο τυπικής απόκλησης ή αν θέλετε διαφοροποίησης ό,τι αφορά τον πληθωρισμό μεταξύ των διαφόρων 14 ε, ε, περιοχών στατιστικά και της Ευρωζώνης. Έχουμε την ίδια τυπική απόκληση για την ανάπτυξη. Κάτι ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι έχουμε την ίδια ε, εξέλιξη στο μοναδιό εργασιακό κόστος και έτσι έχουμε ανταγωνιστικότητα με τους ενδιαφόρων πολιτιών και μοιάζει ε, το σχήμα αυτό της εξέλιξης στο κόστος του εργασιακό, μοιάζει με το κόστος στην Ευρωζώνη. Έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Αλλά έχουμε και τεράστιες διαφορές. Παραδείγματο χάρη απασχόληση ανεργία. 13,5 άντε 14% είναι το υψηλότερο ποσοστό ανεργία στη ΣΥΠΑ και το χαμηλότερο 3,4 με 3,5. Αυτή είναι η απόσταση. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Όταν κάποιος έχει να χειριστεί μια αχανή ενιαία αγορά με ένα ενιονόμισμα πρέπει να περιμένει μεγάλη διαφοροποίηση και πολυμορφία. Πώς τη διαχειρίζεται, αυτό είναι το θέμα. Στη ΣΥΠΑ υπάρχει όμως πανδιακή κυβέρνηση. Στην Ευρώπη πρέπει σίγουρα η διακυβέρνηση να βελτιωθεί. Αυτό είναι προφανές και νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ήδη από σήμερα στο πώς σήμερα ήδη μπορούμε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και τη δημοσιονομική επιτήρηση και εποπτεία, αλλά και την ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Αυτό άλλωστε συζητάτε και εσείς με το Συμβούλιο του Παρόντος. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντλήσουμε τα διδάγματα από την κρίση και θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε αύριο και τι θα κάνουμε μεθαύριο. Έχω πει πρόσφατα σε ομιλία μου ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε αύριο είναι να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να είμαστε σε θέση σε μια χώρα. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί από μόνη της, να μπορεί το κέντρο, αν θέλει, το πυρήνας, να υποκαθιστά τη χώρα σε κάποια, στη λήψη κάποιων αποφάσεων. Όταν κάποιος είναι στην ενιαία αγορά με το ενιαίο νόμισμα, νομίζω ότι αυτό είναι ε, αναγκαίο. Και τώρα τι θα αποφασίσει ε, ο Ευρώπης θα το δούμε. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά ένας νέος ε, τύπος συνομοσπονδίας, ε, ομόσπονδων ε, συγγνώμη, ε, κυρίαρχων κρατών, ίσω είναι κάτι που θα το αποφασίσει μεθαύριο ο λαό τη Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι δική σα απόφαση, όχι δική μου. Δεν έχω την πρόθεση ως Ελληνίδα βουλευτής να σας ε, ρωτήσω κάτι σε σχέση με την ελληνική κρίση. Θα ήθελα ωστόσο να σας ευχαριστήσω διότι πλησιάζει το τέλος ε, της δικής σας θητείας. Θέλω να σας ε, ευχαριστήσω γιατί παίξατε έναν ε, αποφασιστικό ρόλο ευθύς εξ αρχής για την επίλυση της κρίσης αυτής. Πλησιάζει λοιπόν το τέλος της θητείας σας και γι' αυτό θα ήθελα να βασιστώ και να αναφερθώ στα διδάγματα που αντλούμε εμείς και να δούμε για το μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα δίδαγμα το οποίο αντλήσαμε από την κρίση είναι ότι πρέπει να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε και θεσμικά και πολιτικά την Ευρωζώνη. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Το βλέπουμε, καθίσατε σαφέ όλο και περισσότερο. Πώ βλέπετε εσεί την αναγκαιότητα αυτή, παραδείγματο χάρη. Γνωρίζουμε και επαναλαμβάνω με την ευκαιρία αυτό που είπαν συνάδελφοί μου. Έχετε εκφράσει επιφυλάξει σε ό,τι αφορά τα ευρωομόλογα. Βέβαια ταυτόχρονα έχετε αναφέρει ριζοσπαστικέ ιδέες, παραδείγματο χάρη ορισμό ενό ενός Υπουργού Οικονομικών για την Ευρωζώνη. Επομένω, αυτή είναι την αναγκαιότητα για τη θεσμική ενίσχυση και την πολιτική ενίσχυση της Ευρωζώνης. Πώς τη βλέπετε και σε αυτό το ίδιο πλαίσιο. Τι ρόλο βλέπετε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το μέλλον θα πρέπει να περιοριστεί ο ρόλος στη σταθερότητα των τιμών. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό μήπως σε σχέση με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και αν ναι, αν υπάρχει κενό, πώς μπορούμε να το γεμίσουμε, να το καλύψουμε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας καταρχήν. Για να ξεκινήσω από την τελευταία σας ερώτηση. Εμείς πιστεύουμε ότι το να δώσουμε στην έκμη σταθερότητα των τιμών, όπως ορίστηκε η συνθήκη, είναι ο ορθός τρόπος ε, για να δώσουμε στην Ευρωζώνη μια άγκυρα σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Αυτό είναι απαραίτητο, θεμελιώδη. Θεωρούμε ότι είναι ένα δεδομένο. Βρισκόμαστε σε μια σταθερή ζώνη με σταθερότητα των ε, τιμών ε, σε επίπεδο 331 εκατομμυρίων κατοίκων ε, τη ε, περιοχή αυτή. Αυτό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη των συμπολιτών μα, Έτσι λοιπόν, ε, μιλώ για όλου του πολίτε των 17 χωρών. Πρόκειται και επίσης και για θεμελιώδη εμπιστοσύνη απέναντι στον ε, υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή η εμπιστοσύνη των επενδυτών ε, και ε, όσων μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσει εργασία στην Ευρωζώνη. Θα σας δώσω μία ένδειξη που νομίζω δεν είναι πολύ γνωστή από την τη δημιουργία της Ευρωζώνης. Δημιουργήσαμε στην Ευρωζώνη 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, καθαρά για να συγκρίνουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε 8 εκατομμύρια καθαρές θέσεις εργασίας στη ΣΥΠΑ. Έτσι λοιπόν, για δύο ζώνες που είναι αντίστοιχης, ε, ε, αντίστοιχου μεγέθους, ε, σας δίνω μία ένδειξη για το τι έγινε. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τώρα να ικανοποιηθούμε με αυτό. Χρειάζονται πάρα πολλές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και πάρα πολλή δουλειά για να βελτιωθούν τα πράγματα. Τώρα, για να επανέλθω στην ερώτησή σας ε, για τις βελτιώσεις ε, σε μια μεσοπροθεσμή και πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά σήμερα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συνθήκη, απαιτεί ε, πολλή δουλειά, έτσι λοιπόν θα πρέπει να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, εδώ για το θέμα αυτό έχω δει τοποθετηθεί όταν ε, οι Ευρωπαίοι θα αποφασίσουν ε, και φυσικά είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι λαοί μας αυτές. Ε, δηλαδή οι λαοί στα δημοκρατικά καθεστώτα θα αποφασίσουν τι θα κάνουν αύριο και μεθαύριο. Νομίζω ότι αύριο πρέπει να έχουμε ένα κέντρο ικανό να λαμβάνει πολύ σημαντικές αποφάσεις για κάποια χώρα αν αυτή δεν το καταφέρνει γιατί θα είναι προς το συμφέρον της ενδιαφερόμενης χώρας φυσικά προς το συμφέρον του συνόλου της Ευρωζώνης. Και μεθαύριο πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν αλλά είναι οι λέει που θα αποφασίσουν, μπορούν να αποκτήσουν μια σύνομοσπονδία διαφορετική φυσικά από τις Ηνωμένε Πολιτείε με έναν Υπουργό Οικονομικών για να διαχειρίζεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα θέματα, αλλά φυσικά θα έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για την Ομοσπονδία κυρίαρχων κρατών. Βέβαια δεν θέλω να πάω πιο μακριά γιατί οι λαοί το αποφασίζουν αυτά. Sylvie, you're looking very agitated there. Sylvie, Πολύ σύντομα. Ε, συγγνώμη. Και τελικά σε ποιον θα λογοδοτεί αυτός ο Υπουργός Οικονομικών ε, ο οποίος αναφέρεται. Ε, κοιτάξτε, εγώ ξέρω σε μια δημοκρατία πρέπει να λογοδοτεί το κοινοβούλιο. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε ένα κοινοβούλιο. Μου αρέσει το γερμανικό μοντέλο. Κοιτάξτε, αν έχουμε μια συνομοσπονδία, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, θα έχουμε μια συνομοσπονδία, θα έχουμε μια συνομοσπονδιακή κυβέρνηση και θα είναι φυσικά υπεύθυνη ε, απέναντι και στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω τώρα εδώ να σας αντικαταστήσω. now we'll go back to the official. Ωραία. Πάμε τώρα στον κανονικό μας κατάλογο από το Άλντε, ο Θόδωρος Κλακάκης. Σκυλακάκης. Mr. President, thank you for being here. Πρόεδρε, ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Δυστυχώ θα πρέπει να θέσω ένα ερώτημα για την Ελλάδα, αλλά σημαντικό. Μιλήσατε πολύ για τι ιδιωτικοποιήσει στην Ελλάδα και το σχετικό πακέτο και όντω ε, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει, κάποια, μια, υπάρξει μεγάλο τέτοιο πακέτο ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα. Είναι αρκετά γενναίο το πακέτο αυτό. Αλλά εάν πουλήσουμε όσο υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας. Δεν θα πάρουμε πολύ χαμηλές τιμές για, τους, ε, για αυτά που θα πουλήσουμε, για τα περιουσιακά μας στοιχεία. Και επίσης, εάν α, ε, ε, μια, μια αγορά που, κατα, που καταπίπτει μέσα σε δύο-τρία χρόνια δεν υπάρχει Κίνδυνο να έχουμε πολύ χαμηλά έσοδα από το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση επιπτώσεων για, τους, ε, για τις τιμές που θα υπάρξουν, ε, που θα λάβουμε αν πουλήσουμε τέτοια περιουσιακά στοιχεία και σε ό,τι αφορά τα κράτη που δανείζουν την Ελλάδα. Είναι σοφό να έχουμε πακέτο 2 εκατομμυρίων κάθε εβδομάδα για τα επόμενα 4,5 χρόνια. Και αν πούμε ότι και αν οι πωλήσει δεν προχωρήσουν στο επίπεδο των τιμών που θέλουμε, υπάρχει κάποια εναλλακτική, ένα πλάνο, ένα πλάνο Β με ένα χρονικό περιθώριο ας πούμε 6-7 χρόνων με, που να μας εξασφαλίζει ψηλότερα εισοδήματα. Ευχαριστώ. We are for the Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ε, Ευρωζώνη στο σύνολό της. Μου ζητάτε τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για ευθύνες της δικής σας κυβέρνησης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που επίσης πρέπει να θέσει τους όρους για τη δική του βοήθεια στη δική σας κυβέρνηση και, και την ευθύνη της κυβέρνησής σας να ε, επανακτήσει την αξιοπιστία της. Και βεβαίως έχουμε και την Κομισιόν που παίζει το ρόλο της η Κομισιόν βρίσκεται σε, σύνθεση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν σχεδιάζουμε εμεί το πρόγραμμα, δεν βάζουμε εμείς τις λεπτομέρειες. Αυτό που ελπίζουμε ε, θερμά είναι όλη η Ελλάδα και ο δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα και όλε οι υπόλοιπε κοινωνικέ ομάδε να καταλάβουν ότι εάν από μόνοι του παίξουν το, το παιχνίδι ενό νικητή, θα αλλάξει απόλυτα η εικόνα που υπάρχει. Και σε ό,τι αφορά την παρούσα κατάσταση, εάν ε, δείτε τις χώρες που είχαν ε, μια κατάσταση δραματική να αντιμετωπίσουν, ε, θα δείτε εάν οι ξένες άμεσες επενδύσεις έγιναν περισσότερες μετά από ότι πριν, όσο ζούσαν δηλαδή το δράμα. Πραγματικά σκεφτείτε το, σκεφτείτε ποια παραδείγματα υπάρχουν ως προς αυτό παντού στον κόσμο. Αλλά και πάλι λέω, το πρόβλημα είναι να υπάρξει εμπιστοσύνη. Εάν έχουμε το πρόγραμμα αυτό των, της προσαρμογής, το οποίο θα ακολουθηθεί πολύ προσεκτικά, εάν υπάρχει, αν εφαρμοστεί με πιστικό τρόπο το όλο πρόγραμμα, θα δείτε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ο ρεαλισμός του υπόλοιπου κόσμου, του των υπόλοιπων Ευρωπαίων, των υπόλοιπης Ευρωζώνης, εξαρτάται από, το, από αυτό που βλέπουν. Είναι απλά τα πράγματα. Και βεβαίως ενθαρρύνω όλους όσους έχουν ευθύνη να κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν την ε, εμπιστοσύνη. Ε, ισχύει για την Ελλάδα, ισχύει και για, άλλους, για άλλες χώρες. Και όντως είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες από το 2007-2008 Πρέπει λοιπόν να προσπεράσουμε αυτό το σκόπελο στον οποίο έχουμε βρεθεί. Όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες. Είμαστε σε έναν, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι απαιτητικό, που είναι δύσκολος, που μπορεί όντω να συμβούν και ε, γεγονότα που δεν τα περιμέναμε. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να προστατευτεί κανείς είναι να βρίσκεται μπροστά στο παιχνίδι, όχι να ακολουθεί τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Για το ECR, e <clears throat> Ευχαριστώ. Αυτό το κοινοβούλιο έχει τονίσει την ανάγκη για αυξημένη διαφάνεια και δημοσιοοικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση του κάθε κράτου μέλου και φυσικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και την υποχρέωση λογοδοσία του συλλογισμού και οποιαδήποτε μηχανισμού χρηματοδότηση και όλε τι συνιστώσει που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη για τον προπολογισμό. Πιστεύετε ότι έχει γίνει επαρκή πρόοδο προ αυτή την κατεύθυνση στην ΕΚΤ. Πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι η ευθύνη και η εμπιστοσύνη που θα μπορούσαμε να δούμε να προκύπτει από όλα τα στοιχεία είναι θεμελιώδης και στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ζωτική σημασία. Εμείς καλέσαμε τη Eurostat να είναι πλήρως αμερόληπτη και ανεξάρτητη, να μπορεί να πάει επί τόπου, να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, να έχει την τεκμηρίωση και να προβεί στη δική της έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, αλλά δεν ε, θα έλεγα ότι αρκεί. Θα έλεγα ότι θα είμαστε απόλυτα ηρεμοί, ησυχοί όταν θα έχουμε ένα ευρωπαϊκό όργανο που θα έχει την ε, ικανότητα να τα ψάξει όλες τις διάφορες χώρες και θα μπορεί να είναι αξιόπιστο στα μάτια όλων. Όπως είπαμε, σε αρκετές ε, χώρες εξακολουθεί να υπάρχει πολύ δημόσια συζήτηση μεταξύ κυβερνήσεων και αντιπολίτευσης για το αν είναι σωστά τα νούμερα ή όχι. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Δηλαδή μια δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν υπάρχει τέτοιου είδους διαφωνία. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, παρόλο παρά τις δυσκολίες που έχουν, μας δίνουν ένα παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί κανείς ε, δεν ε, φέρνει αντίρρηση για τα αριθμητικά στοιχεία. Ε, δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοιες διενέξεις για τη σημερινή εικόνα, μπορεί για τις προβολές, ναι, για το μέλλον. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και για τους 17. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Um... Γίτσες, κυρία Πρόεδρε. Ο ε, κύριο Τρισέ θέλω και εγώ να τον ε, συγχαρώ για το βραβείο και το βραβείο Καρλομάγνου. Ε, είναι όντως σημαντικό αυτό που έγινε στο Άχεν, ειδικά αν δούμε και τις συζητήσει που γίνονται σήμερα στη χώρα μας για, την, για το ευρώ. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της αφαιρεγγιότητας της Ελλάδας. Καταρχάς, για μένα δεν είναι εξηγήσιμο πώς μια χώρα στην κατάσταση της Ελλάδας μπορεί να έχει ε, πλεόνασμα 4-5% με τέτοια ύφεση. Μιλάτε για ιδιωτικοποιήσεις, αλλά ο συνάδελφος πριν από μένα είπε ότι όταν κάποιος ιδιωτικοποιήσει κάτω από πίεση δεν πετυχαίνει καλές τιμές και γεγονός είναι ότι μάλλον υπάρχει έτσι μια μεγάλη πίεση για να ιδιωτικοποιήσει και δεν επιτυχάνει τελικά αυτά που είχε ελπίσει να επιτύχει. Η ιδιωτικοποίηση λέτε ότι έχει κάποια πλεονεκτήματα και για οικονομικούς λόγους. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά όταν κάποιος πουλάει κάτω από πίεση, δεν παίρνει αυτή την ελάφρυνση ε, στην, στο χρέος του που θα έλπιζε. Είναι μεγάλη λοιπόν η, η πίεση, ακριβώς λόγω του υψηλού κρατικού χρέους. Και αυτή δεν μπορούμε να την, έτσι, να την αποφύγουμε. Και η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων κάτω από τέτοια πίεση δεν θα είναι τόσο αποδοτική. Προφανώς θα καταλήξει και σε απώλεια της κρατικής περιουσίας σε παράλογες τιμές. Είπατε και για την Ασία. Στην Ασία, στην Νότια Κορέα και στην Ταϊλάνδη αναδιαρθρώθηκε ένα κομμάτι του χρέους και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πρέπει να, θα ήθελα μάλλον να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Γιατί δεν είναι αυτή μια κρίση φερεγγιότητας. Και επίσης θα ήθελα αν, να μου πείτε, αν μιλούμε για εθελοντική ε, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα δικά της ομόλογα και τα δικά της, τη δική της κατοχή σε ομόλογα, θα συμβάλλει και αυτή εθελοντικά για να μειωθεί η κρίση φερεγγιότητας που υπάρχει στην Ελλάδα. Again, I, uh, would expect, uh, if I may... Uh, Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ε, περίμενα να έχω κάποιες ε, ερωτήσεις για την νομισματική πολιτική, το επίπεδο του πληθωρισμού, πώς θα είναι ο πληθωρισμός σε δύο χρόνια, αν οι προβολές μας είναι σωστές ή διασφαλμένες και αν έχουμε τα ε, σωστά επιτόκια λαμβάνοντας υπόψη και αποφάσεις που λαμβάνονται σε άλλα μέρη του κόσμου. Αλλά βλέπω ότι έχετε τέτοια εμπιστοσύνη στην τράπεζα που ούτε καν σας απασχολεί αυτό. Δεν το θεωρείτε καθόλου πρόβλημα. Και έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για θέματα που δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για την Ευρωζώνη συνολικά, τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη συνολικά. Το λέω και το ξαναλέω αυτό. Τώρα, αν έχουμε ένα μόνιμο και γενικό διάλογο, συζήτηση, γιατί όλα αφορούν ε, το γενικό ενδιαφέρον, είναι ένα γενικό ε, θέμα Είμαστε στο επίκεντρο παγκόσμιων γενικών ε, εντάσεων και έχουμε παγκόσμιους κινδύνους να αντιμετωπίσουμε. Αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να επανέλθω τώρα σε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, από το υψηλό επίπεδο κατανόησης να περάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο, σε ένα χαμηλό μάλλον, ξέρετε τι έγινε και τι έγινε στο Βέλγιο. Από το 135 στο 85. γιατί είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιμονή και ακολουθούσαν μια πολιτική που οδήγησε σε ανάπτυξη και σε δημιουργία θέσεων εργασίας, σε εξυγίανση, σε σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα. So to run policies without the... Αν δεν υπάρχει η ε, λοιπόν ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δούνου του, το λεγόμενο αυτό conditionality, αιρεσιμότητα και αν δεν υπάρχουν και όλες αυτές οι άλλες, ναι αυτό θα ήταν πιθανό. Θα μπορούσα να αναφέρω την Ιταλία. Γνωρίζουν οι Ιταλοί που είναι σήμερα εδώ παρόντες ότι έχει γίνει εκπληκτική προσπάθεια τη δεκαετία του 90. Δεύτερον, για τις ιδιωτικοποίησεις τα είπα, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Η κυβέρνηση αποφάσισε να προβεί σε ιδιωτικοποίησεις και νομίζουμε ότι η απόφασή της ήταν πάρα πολύ σημαντική και πολύ σωστή. Τώρα, το πώς θα βελτιστοποιηθούν οι ιδιωτικοποίησεις είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. αλλά οι αρμόδιοι θα το διαχειριστούν. Τα κατάλληλα άτομα θα το διαχειριστούν. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό για τη μακροχρόνια αξιοπιστία μιας χώρας. Κάτι που δεν ισχύει για τις περισσότερες άλλες χώρες. Πρέπει ε, να ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αναζωογόνηση και ενίσχυση της οικονομίας της χώρας. Τώρα, κατά τα λοιπά, να επαναλάβω ότι αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστικότητα της ίδιας της χώρας. Στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησής της και των πολιτικών ευαισθησιών. Παρακολουθούμε τι γίνεται στην ε, Ελλάδα. Ξέρουμε ότι έχει μια παγκόσμια εμβέλεια θα έχει επιπτώσει παγκόσμιο επίπεδο και θα δούμε και εμείς πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την κατάσταση. Εμείς από τη δική μας πλευρά παρέχουμε συμβουλές στους αρμόδιους να λάβουν τις αποφάσεις. Δεν τους αντικαθιστούμε αυτούς. Δεν μπαίνουμε στη θέση τους. Η δική μας εντολή είναι να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών για 331 εκατομμύρια άτομα. Λίγο λιγότερο από ό,τι ο πληθυσμό των ΗΠΑ. Uh, Συγγνώμη, δεν μου απαντήσατε στην ερώτησή μου για το αν θα συνεισφέρετε σε αυτές τις εκούσιες προσπάθειες, την εκούσια διακράτηση ε, των ομολόγων. Ε, κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όχι του δημόσιου τομέα και έχω πει ήδη ότι εμείς δεν σκεφτόμαστε να συμμετάσχουμε. Μάλιστα, αυτό είναι ο νομισματικός διάλογος ε, και όχι ο συμβουλευτικός διάλογος. Το θέμα είναι ότι εσείς ε, δεν είστε υπεύθυνο για κάποια πράγματα, αλλά θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας, ε, γιατί σεβόμαστε την απόψή σας. Λοιπόν, για το ΕΛΚ, κύριο Λένιν. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, αγοράστηκαν ούτως ή ε, ο ομόλογα από την δευτερογενή αγορά. Ε, άκουσα, διάβασα χτες μάλλον ότι είχαν, είχαν στόχο την ρευστότητα αυτή που τα αγόρασαν. μιλήσατε πριν για ένα κβαντικό και, άλμα. Ε, το ένα ε, το άλμα αυτό σημαίνει ότι κάποιο θέλει να πηδήξει. Το Συμβούλιο βλέπουμε ότι είναι με το ένα πόδι στη γη. Δεν θέλει να πηδήξει, δεν θέλει να το κάνει το άλμα. Ε, εσείς τι μα συμβουλεύετε αν το Συμβούλιο συνεχίσει να μπλοκάρει. Το Συμβούλιο έχει στυλώσει τα πόδια και υποστηρίζεται από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτή την πρόοδο λοιπόν που έχουμε κάνει, τι θα την αναβάλουμε για το μέλλον και μπορεί να διακινδυνεύσουμε ας πούμε οι σοσιαλιστές να μην να συμπράξουν ή θα πρέπει να οξύνουμε το, ή να, θα πρέπει να απαλύνουμε μάλλον το α, πακέτο σταθερότητα και ανάπτυξη. Ε, ναι, τη γνώμη του θέλω, τη γνώμη του θέλω. Και το τρίτο, γίνονται και κάποια σχόλια εκτός μικροφώνου, ο τομέας των τραπεζών έχει ένα, πλάνο δεύτερο, ένα δεύτερο πλάνο για την Ελλάδα. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ή, να δώσουμε στην Ελλάδα την ευθύνη που της αναλογεί. Αλλά θυμάμαι ότι πριν από ένα χρόνο μιλούσαμε για ε, ε της, ε, ε, της Ευρωζώνης και κανένας δεν ήθελε πλάνο, δεύτερο πλάνο, δεύτερο σχέδιο. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει κάποιος, το έχει κάποιος. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο πλάνο. Δεν μπορώ να με φανταστώ δηλαδή ότι η συζήτηση γίνεται μόνο με το, με το πρώτο σχέδιο και δεν υπάρχει θέση αναδίπλωσης. Βεβαίω, δράτω ε, και τι ευκαιρίε να σα ε, συγχαρώ για την ε, έκτηση τη θητεία σα, παρόλο που είχατε κι εσεί αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και η Ευρωπαϊκή Κρατική, Κεντρική Τράπεζα σας ευχαριστεί. Για το πρώτο που είπατε. Επαναπορροφήσαμε την ρευστότητα που είχαμε δώσει μέσω του S&P κάθε αναβδομάδα. Οπότε δεν προσπαθούμε να αποσκοτικοποιήσουμε τα πράγματα. Απλώς απορροφήσαμε την α, ρευστότητα που υπήρχε. Τώρα, για αυτό το κουβαντικό άλμα. Είναι σαφές το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Κεντρικής Τράπεζας για το τι προτείνουμε να κάνει η Ευρώπη. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Δεν είμαστε εμείς καν στον τριμερή διάλογο. Εσείς είσαστε. Και οι κυβερνήσεις των ε, κρατών και οι κομισιόν. Όχι γιατί κάποιες χώρες βρίσκονται σε μια αλφα κατάσταση, κατά αναγκή, έχουν και δίκιο. Το έχουμε δίκιο στο παρελθόν αυτό. Ας πούμε για το πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξης και ξέρουμε ότι τώρα, ε, εκ των υστέρων, μπορούμε να δούμε ότι δεν ήταν τελικά σωστό να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τούτου λεχθέντος, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Εμείς απλώς λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον βέλτιστο βαθμό για να βελτιώσουμε την ε, διακυβέρνηση. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω ότι είναι πολύ περίπλοκο και να πω επίσης, επειδή το αναφέρατε, ε, ότι υπάρχουν έτσι αρκετές ευαισθησίες, εμείς εκδίδουμε ε, το νόμισμα για όλους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολυεθνική και με πολλές ευαισθησίες. Μας αφορούν όλοι οι πολίτες όταν παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Ε, σχέδιο αναδίπλωσης. Αυτό που κάνουμε είναι ένα εγχείρημα, όχι για την α ή τη β χώρα ή τη γ ή τη δ ή την ε, ή για την ε, Ευρωζώνη ή για την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα παγκόσμιο. Και αυτό θέλω να το πω σαφώς. Συζητούμε έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία για κάτι που ουσιαστικά είναι η πρώτη χρεοκοπία μιας ε, προηγμένης χώρας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε και πάλι νομίζω ότι πρέπει να, είμαστε, να δείξουμε την απαραίτητη ευθύνη. Και σε ό,τι μας αφορά, εμείς επαγρυπνούμε πάντα. Έχουμε αυτή την έννοια της μόνιμης επαγρύπνησης. Θα θυμάστε ότι όταν ξεκίνησαν οι αναταράξεις στην 9 Αυγούστου 2007 πήραμε την πρώτη πολύ σημαντική απόφαση. Μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε είμαστε μόνιμα σε επαγρύπνηση και μπορείτε να βασίζεστε σε αυτή την επαγρύπνηση αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι το επίπεδο ευθύνης από αυτούς που είναι στην εξουσία, δηλαδή από τις κυβερνήσεις. Και βεβαίως και από τη διεθνή κοινότητα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την Ευρώπη την οποία εκπροσωπεί σε αυτόν τον τριμερή διάλογο η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές ο Ρόμπερτ. Πρόεδρε. Εδώ και δύο χρόνια η Ελλάδα είναι σε ύφεση και το ΕΕΠ συρρυκνώνεται και φυσικά αυξάνεται, διωγγώνεται συνέχεια το χρέος σε σχέση με το ΕΕΠ. Το πακέτο βοήθειας ε, του Διεθνούς Ομοσπονδίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι πρόσθετο χρέος ε, τελικά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το επιτόκιο, πολύ μεγάλο το επιτόκιο μια πραγματικά ευρωπαϊκή λύση θα ήταν να δημιουργηθεί μια ε, ολοκληρωμένη αγορά. Ε, σας τέθηκε αυτή η ερώτηση από συναδέλφους, αλλά δεν απαντήσατε. Ε, μια ε, τέτοια αγορά ήδη θα μπορούσε να υπάρχει. Υπάρχουν ε, ήδη και τα ευρωμόλογα ή έκτε με την εγγύηση των 27 τα εξέδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ αξία για με ένα επιτόκιο 4% κάτι τέτοιο θα επέτρεπε σε όλες τις κυβερνήσεις να επαναχρηματοδοτηθούν και να βρουν το δρόμο της δημοσιονομικής αιρετής και να επενδύσουν εκ νέου. Εσείς δεν θέλετε χρεοκοπία, ε, αλλά γιατί δεν υποστηρίζετε αυτή την ιδέα που ε, πρόθεσαν οι κύριοι Γιουκέρ και Τρεμόντι και το Ινστιτούτο Μπρέγκελ. Ε, νομίζω ότι θα ήταν ε, μία οδός που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρώπη να βρει μία μεγαλύτερη ενότητα και κατόπιν να αναδιαρθρωθεί. Και για να κλείσω, επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ ήρεμες διακοπές, χωρίς κρίση. Στην περιοχή που και οι δύο αγαπάμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την τελευταία σας ευχή και χαίρομαι που και εμάς μας αρέσει το ίδιο μέρος για τις διακοπέ. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση που θέτεται είναι πραγματικό ζήτημα. Η θέση του Συμβουλίου ε, των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων τη στιγμή που μιλώ είναι ότι, όπως έχω ήδη πει, ζητήσαμε το μέγιστο επίπεδο ευελιξίας για το EFSF ε, και για το ESM. Το EFSF είναι σήμερα, η ESM θα μετατραπεί αύριο, θα μετατραπεί στο μηχανισμό αυτό. Και πρόκειται για ένα μέσο που, όπως ξέρετε, αναχρηματοδοτείται ε, από την αγορά με πολύπλοκες εγγύησεις, αλλά αυτές καθορίζονται από κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε το μηχανισμό το σταθερότητα σήμερα και αύριο του ESM. Ξέρετε ότι ε, εδώ θέλουμε τη μέγιστη ευελιξία, αλλά πρέπει να δούμε και το θέμα της ερεσιμότητας της πολλαπλής συμμόρφωσης. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα αυτό, κατά τη γνώμη μας. Ευχαριστώ πολύ, Ραμόν, για τους φιλελευθέρους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, η ΕΚΤΑ διαδραματίζει και έναν φορολογικό ρόλο, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά και το δημόσιο χρέο. Για να μην έχει αυτό το ρόλο η ΕΚΤΑ, μήπω θα ήταν αποτελεσματικό και χρήσιμο να υπάρχει όχι μόνο ένα Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών, αλλά και ένα ε, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών. Και ένα δεύτερο πολύ σύντομο ερώτημα. Σας ανησυχεί ο συντελεστής μόχλευσης της έκτης. Στα τέλη του 2010 μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ ενεργητικού και αποθεματικού, ε, είχαμε ένα 24, ενώ σε άλλες ε, χώρες ε, αυτό το leverage ratio, αυτή, αυτός ο λόγος μόχλευσης, είναι γύρω στο 4 με 6. Στη Lehman Brothers ήταν 30. Σας ανησυχεί λοιπόν αυτό το νούμερο. We, we have a tendency... Εμείς έχουμε την τάση να συγκρίνουμε την Ευρώπη με τη ΣΥΠΑ, αλλά και άλλες σημαντικές κεντρικές τράπεζες παρόμοιου μεγέθους. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοια μεγέθη και παρόμοια συμβάντα. Αν δει κανείς τον ισολογισμό του ευρωσυστήματος αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες, στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις που έχουμε, στα πιο πρόσφατα στοιχεία και αν αυτά τα στοιχεία τα συγκρίνουμε προ, με τα πρώτης κρίσης στοιχεία, τέλη Ιουνίου 2007, σε ό,τι αφορά λοιπόν το μέγεθος του συνολικού ισολογισμού, είχαμε αύξηση της τάξης των 600 δις. Από 913 πήγαμε σε 1,5-3 περίπου. Άρα μιλάμε 1,7 κατά μία φορά, κατά 1,7 αύξηση. Και έχει και να κάνει αυτό και με την τιμή του χρυσού βέβαια. Αλλά και άλλα φαινόμενα που έπαιξαν εκείνη την εποχή ρόλο. Αν επικεντρωθώ στην νομισματική πολιτική, τα μέσα νομισματικής πολιτικής, βλέπω εδώ αύξηση πολύ πιο μετριοπαθή. Κατά 20% περίπου. Τώρα, αν συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τις ΙΠΑ, είναι μια φυσική σύγκριση αυτή, από 845 δις δολάρια πριν την κρίση πήγαμε σε 2,75-3. Τριπλασιασμός δηλαδή στην περίοδο αυτή. Λίγο παραπάνω, μάλιστα. Άρα, ναι μεν έχουμε αύξηση συνολικά του ισολογισμού μας, αλλά είναι πιο μετριοπαθής αυτή η αύξηση. Ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα αντίστοιχο σύστημα με την ε, Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε ό,τι αφορά το μέγεθος και την ε, αύξηση συνολικά του ισολογισμού. Πάντω και εμεί είδαμε σημαντικές αυξήσει και των αποθεμάτων και ε, σε χρυσό συγκεκριμένα. Να σας πω ότι προσέχουμε πάρα πολύ ό,τι κάνουμε. Έχουμε ένα πλαίσιο όπως σας είπα για τις εγγύσεις συνολικά τα collaterals. Προσπαθούμε να είμαστε στο δυνατόν πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που αναλαμβάνουμε τα ρίσκα που παίρνουμε και μία μόνιμη μέρημνα και ανησυχία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ακριβώς αυτή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κάνουμε αυστηρά, όπως σας είπα, τη διάκριση μεταξύ των πρότυπων και μη πρότυπων μέτρων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, διότι θα πρέπει να παραδώσω τη σκητάλη της Προεδρίας στον Αντιπρόεδρο, διότι όπως σας προείπα πρέπει να προεδρεύσω του τριμερούς διαλόγου για την οικονομική διακυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλετε να είμαι εκεί και όχι εδώ. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι δεν είναι η τελευταία φορά που έχουμε μαζί μας ε, τον ε, κύριο Τρισέ. Θα μας ξαναεπισκεφτείτε και στις 19 Σεπτεμβρίου, κύριε Τρισέ. Θέλω όμως και εγώ, όπως και όλοι οι πολλοί προλαλήσαντες, να εκφράσω την ε, εκτίμησή μου για το έργο που έχετε επιτελέσει μέχρι τώρα. Θα με αντικαταστήσει λοιπόν αντιπρόεδρος. Έχετε ε, νομίζω πέντε ακόμη ομιλητές, αλλά τέλος πάντων ο αντιπρόεδρος αντικαταστήσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Παρακαλώ λοιπόν να είστε όλοι πάρα πολύ σύντομοι σε ερωτήσεις σας. Κυρία Άστριντ Λούλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και αν δεν είναι η τελευταία σας ακρόαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ακούραστε προσπάθειες που καταβάλατε κατά τη διάρκεια τη θητείας σα και κατά τη διάρκεια τη ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης προκειμένου να εγγυηθείτε τη σταθερότητα του ενιαίου μας νομίσματος. Είμαι σίγουρη ότι οι ιστορικοί θα αποτίσουν ε, το φοροτιμής ε, ε, που σας ε, αξίζει γιατί ε, τα συμβάντα των τελευταίων ετών θα είχαν αφήσει πολλούς πολιτικούς άφωνους ή σχεδόν. Έχω μια ερώτηση στο πλαίσιο αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών για το 2020. Η Κομισιόν προτείνει την θέσπιση ενός φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ίδιους πόρους εσείς έχετε κρούσει τον κοδόνα του κινδύνου στο να ληφθεί ένα τέτοιο μέτρο μόνο σε επίπεδο έχει κρουθεί ο κόδωνα του κινδύνου για το να τεθεί ένα τέτοιο μέτρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Εσείς τι πιστεύετε για την πρόταση αυτή, η Κομισιόν πιστεύει ότι τα έσοδα θα είναι από 30 έως 50 ε, δισεκατομμύρια. Είναι ρεαλιστικό ή είναι λαϊκιστικό, όπως πιστεύουν ορισμένοι, γιατί θέλει η Κομισιόν τώρα να αποδείξει ότι ποινικοποιεί τη τράπεζες ε, και θα πρέπει ε, να έχουμε φορολογικά έσοδα μέσω του ποινικού δικαίου και θέλω να μου πείτε και κάτι για το μηχανισμό, μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων που αν εγκριθεί από τα κράτη-μέλη θα αρχίσει να ισχύει από το 2013, από τον Ιούνιο του 2013. Τι πιστεύετε για την αγορά των ομολόγων ε, των κρατών μελών της Ευρωζώνης ε, στην αγορά. Ε, δεύτερον, για τη δυνατότητα ο μηχανισμός αυτός να δίνει εγγυήσει αντί για τις κρατικές εγγυήσει. Τρίτον, τι πιστεύετε για την νομική φύση αυτού του μηχανισμού και για την ενδυνάμει επεκτασή του. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν θα σας εξεπλήξει η απάντησή μου για την πρώτη ερώτησή σας. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ένας ειδικό όρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που θα επιβαλλόταν στην Ευρώπη και δεν θα ίσχυε στον υπόλοιπο κόσμο και μάλιστα στα κύρια χρηματιστήρια, στις κύριες αγορές θα σήμαινε σημαντική απώλεια δραστηριότητα για την Ευρώπη και έτσι λοιπόν ε, θα είχαμε τέτοιες αρνητικές ε, συνέπειες. Ε, έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν σημαντικότερη δραστηριότητα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ρυθμιστούν οι χρηματαγορές, να ελέγχονται, θα πρέπει να ε, μπουν ε, σε ένα περιβάλλον ε, μέγιστης ανθεκτικότητας, όμως αυτός ο τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις περισσότερες βιομηχανοποιημένες αλλά και για τις αναδυόμενες χώρες. Έτσι λοιπόν, εμείς διατηρούμε την ίδια θέση όπως και στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πιθανή ευελιξία του EFSF και ε, του SME πάντοτε έχουμε ζητήσει μεγάλη ευελιξία, πάντοτε αν θέλουμε να διατηρήσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη μας ενδιαφέρει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα που να είναι προσαρμοσμένα στο σήμερα. Ε, φυσικά θα υπάρχει και ισχυρή πολλαπλή συμμόρφωση ε, πιστική πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό θα το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς, αλλά είμαστε υπέροχοι υπέρ ε, της ε, ευελιξίας, ε, είμαστε υπέρ ε, της παρέμβασης στις δευτερογενείς αγορές, όχι στις πρωτογενείς αγορές. Ε, θα μπορούσαμε να παρέμβουμε υπό τη μορφή εγγυήσεων στις δευτερογενείς αγορές. Πάντως πιστεύω ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία. Ευχαριστώ. Να ζητήσω τώρα από την κυρία Φερέρα και τον κύριο Μπούλμαν να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε μια πιο ελεύθερη προοπτική, μπορούμε να δούμε καλύτερα το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη και απέναντι στην πρότασή σας να έχουμε έναν Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης ε, ως πρώτο ε, βήμα σε αυτή την ε, προσέγγιση τίθεται αυτή η πρόταση γιατί σας το επιτρέπει και το γεγονό ότι λίγη θητεία σας όμως φαίνεται να μην είναι ισορροπημένη αυτή η πρόταση από μόνη της δηλαδή αν δούμε στο παρελθόν και αν δούμε την πορεία που ακολουθήσαμε εγώ αναρωτιέμαι, δεν ε, είναι σημαντικό να σκεφτούμε αν μια ευρωζώνη μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει με ένα προϋπολογισμό που ουσιαστικά ε, είναι ίση με την πρώτη πακέτο στήριξης που χρειάστηκε η Ελλάδα για να επιβιώσει. Ε, βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του δολαρίου και τον έχουμε εμείς ένα ισχυρό προϋπολογισμό είναι σημαντικό θέμα. Τα ευρωμόλογα δεν θα ήταν τώρα η κατάλληλη στιγμή να τα σκεφτούμε και να έχουμε πιο διαφορετικέ λύσει στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με δάνεια που θα χορηγούνται με λογικά επιτόκια για με λογικέ Δεν ε, θα μπορούσε να ε, έρθει αυτή τη στιγμή τώρα να λάβουμε μια τέτοια απόφαση και δεν ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου να αναγνωρίσουμε ότι τα περιθώρια ε, της προσερμογής όταν ε, χώρες ανήκουν στην Ευρωζώνη, σε μια νοσομηματική ένωση, ότι αυτά τα περιθώρια είναι πάρα πολύ περιορισμένα σε σχέση με όσα υλοποιούνται και αυτό θίγει ένα άλλο θέμα που πρέπει να επιληθεί. Το πρόβλημα μιας συνολικής προσέγγισης, ε, συμμετρικής ε, ή ασύμμετρης προσέγγισης όπως την αποκαλούμε, αλλά εξακολουθεί να επιζητά επίλυση αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει να συζητηθεί το θέμα του πακέτου της οικονομικής διακυβέρνησης μεταξύ Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι χώρες δεν έχουν τα μέσα να κάνουν τις προσαρμογές, ακόμη και όταν έχουν ανοιχνευτεί διαρθρωτικές ανισορροπίες. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να ε, μπορέσουν τα κράτη να επενεπενδύσουν στην ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, αλλά θα ήθελα να ακούσω την απάντηση της, στην κυρία Φερέρα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, σας ευχαριστώ. Thank you very much for this... Uh, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα σας έλεγα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα σε αυτό που είναι σημαντικό που είναι η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και βέβαια των 27. Και να επικοινωθούμε και στην πρόοδο που πρέπει να γίνει. Εγώ σας είπα ποια είναι η απόψή μας. Βεβαίως θα σκεφτούμε, θα δούμε, εάν δεν, μπορούμε, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει τώρα, η ιστορία θα μας κρίνει ότι μάλλον ήμασταν πολύ δειλοί. Τώρα για τα ευρωμόλογα είπα ποια είναι η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε την απόφαση να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, το οποίο σήμερα το λένε Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και αύριο θα το λένε ESM. Ένα ταμείο λοιπόν που θα είναι ένα μηχανισμό δηλαδή σταθερότητας, που θα είναι ένα μεγάλο ευρύ ταμείο το οποίο βεβαίως θα την χάνει και τις υποστήριξη του Δονοτού και θα ζητούμε την ε, μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για το Ταμείο αυτό, εφόσον βεβαίως υπάρχει ισχυρίου, υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθεροί όροι. Βεβαίως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά όσοι συμπεριφέρονται σωστά έχουν προφανώ τελείω διαφορετική μεταχείριση από αυτού που δεν συμπεριφέρονται σωστά. Αυτό ισχύει και για την Ευρώπη, ισχύει και για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε τέτοιε καταστάσει. Ισχύει και για τα επιτόκια. Ισχύει και για το δυναμικό ανάπτυξη. Ισχύει και για την αντιμετώπιση τη ανεργία. Κάποιε πολιτικέ και οι απαραίτητε διαρθρωτικέ αλλαγέ προφανώς έχουν και αποτελέσματα, που είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασία. Οπότε εμεί πρέπει να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε κάθε ενέργεια προ αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίω να προλάβουμε την ε, εμπλοκή σε, λανθασμένους, ε, σε λανθασμένες δράσεις, προσανατολισμούς, φορολογικές, πολιτικές. Επίσης, οι δείκτες ανταγωνιστικότητας είναι κάτι πολύ ουσιαστικό Οπότε συμφωνώ ότι είναι απόλυτα θεμητό αυτό που λέτε, αλλά εμείς θα εμείνουμε στην, στη σημερινή μας θέση. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούλμαν, θέλετε το λόγο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Είμαι ο τελευταίος, έτσι δεν είναι. Οπότε να ακολουθήσουμε τον κατάλογο, Πρόεδρε. Αν έχω εγώ το λόγο, εντάξει. Πρόεδρε, ένα ερώτημα έχει παραμείνει ε, κρεμές, που είπε η συνάδελφος, που ανέφερε η συνάδελφος Βάλτς για, τις, ε, για, τις, για τους οίκους αξιολόγησης. Εσείς πόσο ε, ικανοποιημένο είσαστε με την νομοθεσία σχετικά με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε, όπως ρώτησε και η συνάδελφος, ότι για τους ε, οίκους αξιολόγησης υπάρχουν προβλήματα διαστρέβλωσης της αγοράς. Okay, schlecht zu verstehen. Μ' ακούτε, μπορώ να ξαναξεκινήσω, αν, αν, επιτρέπετε. Ωραία. Ήμουνα σε λάθο μικρόφωνο, συγγνώμη. Ήθελα απλώ να επαναλάβω την ε, ε, ερώτηση της συναδέλφου για του οίκου αξιολόγηση. Πόσο ικανοποιημένο είσαστε με την εφαρμογή της νομοθεσίας έτσι όπως την έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο υπάρχουν, τι πρέπει να κάνουμε με τις ε, αν πρέπει να επιμειώσουμε την επίδραση που έχουν και κατά πόσο μπορούμε να προλάβουμε τις επιπτώσεις που είναι διαστρεβλωτικές για την αγορά και απορρέουν από τους οίκους αυτούς. Επίσης, τι πιστεύετε για τους παίκτες κλειδιά στην αγορά. Μιλήσαμε για σταθερότητα τιμών, Μιλήσαμε, για, μιλήσατε για την συμπεριφορά κρατών, μιλήσαμε για την συγκράτηση του πληθωρισμού και ότι κάθε χώρα πρέπει να κάνει το, ό,τι της αναλογεί για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό Σύμφωνα με τη δική σας οικονομική προσέγγιση υπάρχει πρόβλημα αν μια χώρα είναι μονίμως κάτω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πληθωρισμό. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς το βλέπετε. Μια χώρα δηλαδή, ίσως οικονομικά δυνατή χώρα, παραμένει κάτω από το στόχο. Δεν επιτυγχάνει το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον πληθωρισμό. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην ιστορική αγορά. Αποτελεί πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο σας ερώτημα να πω ότι εξακολουθεί το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό θέμα αυτό να είναι ακόμη ανοιχτό. Και πράγματι είπατε ε, ότι το έθεσε και ο συνάδελφός σας. Είναι γενικότερο το θέμα, παγκόσμιο. Προσπαθούμε να είναι λιγότερο προκυκλικός ο κόσμος και τα παγκόσμια οικονομικά. Να μην έχουμε όλες αυτές τις ανακατατάξεις, ε, αυτά τα, τα πάνω κάτω. Και υπάρχουν αυτές οι ευθύοι και αξιολόγησης που είναι λίγοι και έτσι έχουμε μια συγκέντρωση επιρροής. Και όλα αυτά οδήγησαν σε αυτά τα προκυκλικά στοιχεία που είπα κατά το παρελθόν. Βέβαια, ε, έχει επιτελεστεί πρόοδος πρέπει να πω στην κατεύθυνση να αποφύγουμε συγκρούσεις συμφερόντων εντός αυτών των οργανισμών. Βελτιώνουμε την εποπτεία και την επιτήρηση. εν του Ατλαντικού. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα αυτού του ολιγοπολίου, της ολιγοπολιστικής ομάδας εικόνα αξιολόγησης προκυκλικού χαρακτήρα. Αλλά έχουμε ένα γενικό μήνυμα προς όλους τους επενδυτές, μετέχοντες αγορές, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κτλ. Όλοι αυτοί πρέπει από μόνοι τους να μελετήσουν την κατάσταση, να δουν ε, σε τι κεφάλαια επενδύουν, σε τι εταιρείε επενδύουν και όταν οι ρυθμιστές προσπαθούν να αποσπάσουν τους κανόνες ε, κυριαρχίας ή ρυθμιστικούς από τους οίκους αξιολόγησης, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτό, Το να προτείνουμε να δημιουργηθούν νέοι και αξιολόγησεις για να διευρυνθεί το πεδίο είναι και αυτό ανοιχτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, θα ήταν πολύ αυστηρό κάτι τέτοιο, αλλά θα ήταν και αφελές να υποθέσουμε ότι ήδη έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Αυτή είναι η απάντησή μου. Εμέσως υπονοήσατε κάποια χώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε για ποια χώρα μιλάτε. Λοιπόν, θα σας πω τι πιστεύω εγώ. Αν μακροπρόθεσμα κάθε χώρα. Εκτός από πολύ ειδικέ περιπτώσεις. Έχει κάποιες δεκιμάνσεις. Κοντά στο 2%, λίγο κάτω από το 2%, το πολύ 2. Αυτό είναι το όριο αναφοράς. Και το έχουμε προαναγγείλει, αλλά το έχουμε και επιβεβαιώσει και είναι και ένα όριο το οποίο εμπιστεύονται και οι παρατηρητές πολύ σωστά ως κανόνα για τα επόμενα 10 χρόνια. Η Γερμανία, γιατί για τη χώρα αυτή μιλάω, ήταν σε μια ειδική κατάσταση γιατί έπρεπε να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη ε, ήταν σε ε, έλλειμμα όταν ξεκίνησε το ευρώ η Γερμανία. Είναι περίεργο να το λέμε αυτό σήμερα, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα τότε και στο δημοσιοτομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυθόρμητα οι εταιρείε και οι κοινωνικοί εταίροι έκαναν αυτό το οποίο έκριναν ότι είναι απαραίτητο για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν πολύ μικρή εξέλιξη με το μοναδίο εργασιακό κόστος. Υπάρχει εφημερία, υπάρχουν εξαγωγές στη Γερμανία, υπάρχουν θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Πάρα πολύ καλό παράδειγμα λοιπόν αυτό που δείχνει ότι όταν κάποιο συμπεριφέρεται με τον πλέον ε, ορθό τρόπο ανταμείβεται. Από εκεί και πέρα τώρα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο πολύ να έχουμε μία διακύμανση γύρω από το πρότυπο, τον κανόνα θα έλεγα, το μέσο όρο για την Ευρωζώνη, όπως και κατά το παρελθόν, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα 12 χρόνια του ευρώ είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σταθερότητα των τιμών για τη Γερμανία. Παρά το ότι ανέβηκε ε, ΦΠΑ ε, στο 3%. Δηλαδή το ΦΠΑ ήταν κατά μέσο όρο 1,5%. Έτσι λοιπόν ε, δεν πιστεύω ότι αυτό το μονιμό καθεστώς είναι αυτό που λέμε εμείς σταθερότητα των τιμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος τομασμάν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, εμείς ε, στο, στις επιθέσεις, ε, μάλλον στις, στους, στους αγώνες του γενικού ποδοσφαίρου στην Φραγκφούρτη είδαμε πραγματικά να συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα δικαίως κερδίσατε το βραβείο Καρλομάγνου μετά από την δράση σας ως προς αυτό. Τώρα, εγώ προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται με τον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος ε, μας έχει αφήσει πάρα πολύ καλή εικόνα εδώ στην ε, ΕΚΟΝ. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως να πιέζουμε για την επίτευξη των στόχων μας. Και βεβαίως η κατάρρευση της Ένωσης θα πρέπει να αποφευθεί. Αυτό το συνυπογράφετε κι εσείς. Αλλά η συμμετοχή των ιδιωτικών επενδυτών στις ελληνικές εταιρείες θα μπορούσε να είναι μια πιθανότητα αντί για μια εναλλακτική σε, όλη αυτή την, σε όλο αυτό το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Και εκεί υπάρχουν διάφορες θέσεις και αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ο, ο φόρος των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και θα πρέπει να υπάρξει ένα εργαλείο το οποίο να μπορέσει να ε, συγκρατήσει όσους δεν παίζουν με τους όρους του παιχνιδιού. Συμφωνείτε σε κάτι τέτοιο ή θα μπορέσετε ίσως να μας πείτε ποια είναι η στοχοθέτησή σας. Πραγματικά ήταν μεγάλη ευκαιρία σήμερα που ήρθατε εδώ και έχουμε ευτυχώς ακόμα την ευκαιρία να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όσα κάνατε για την ε, Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Να πω απλά ότι δύο πράγματα θέλω να πω για τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Να πω καταρχάς ότι είναι κάτι πολύ ελκυστικό για πολλούς παρατηρητές. Εισήχθη ως ιδέα από τον καθηγητή Τόμπιν που είναι πραγματικά μεγάλο μυαλό, ο οποίος είπε ότι δεν θα προωθούσε κατά ανάγκη έναν Tobin tax σήμερα, έναν φόρο Tobin, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε και τα εξή. Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη γενική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι σωστό να έτσι να ωρεοποιήσουμε λιγάκι την, ε, την κατάσταση, αν δεν λειτουργεί, μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό που δεν λειτουργεί άμεσα. Όχι απλώς ε, να προσπαθούμε να, έτσι, να χτενίζουμε τα πράγματα και να μην αφήνουμε τα συστήματα να λειτουργούν ε, απρόσκοπτα. Επίσης το θέμα της ανταγωνιστικότητας το οποίο είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Εάν κάποιες ε, συναλλαγές θεωρούνται πιο δαπανηρές στην Ευρώπη από, από αλλού στον κόσμο, τότε θα πάνε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, γιατί μπορεί να δει κανεί πώς η παγκόσμια αγορά ομολόγων, ευρωμολόγων πέρασε από την ε, Νέα Υόρκη στο Λονδίνο, ακριβώς επειδή υπήρχε φορολόγηση που δημιουργούσε προς κόμματα ή δημιουργούσε πιο δαπανηρές, ε, έκανε πιο δαπανηρές τις ε, συναλλαγές στη Νέα Υόρκη. Αυτά λοιπόν είναι πραγματικά προβλήματα. Και αν κάνουμε κάτι που δεν είναι οργανωμένο σε, ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό ισχύει για, τις, για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά στον, παρούς, στον παρόντα κόσμο, όπου δεν έχουμε μόνο μια ανεπτυγμένη οικονομία, αλλά έχουμε και τον αναδυόμενο κόσμο, ο οποίος παίρνει τη θέση του, σε κάποιε περιπτώσει, εγώ όταν βρίσκομαι σε τέτοιε χώρε, έχω την εντύπωση ότι αυτοί είναι πολύ πιο πλούσιοι, είναι πιο, πολύ πιο πλούσιε κοινωνίε και οικονομίε από την Δυτική Ευρώπη, α πούμε, ή την Ευρώπη στο σύνολό τη και τη είπα. Πραγματικά λοιπόν ο κόσμο αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και θα ήθελα να ζητήσω μεγάλη σύνεση στο πώς θα προχωρήσουμε. Ξέρετε ποια είναι η θέση μας. Λυπάμαι που δεν πάω προς αυτό που λέτε, δεν κινούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει. Γίνεται όλο και πιο σαφές. Και δεν είναι μόνο αυτό ο τομέα που λέμε ας δούμε τη γενική εικόνα. Ας είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε κάτι που θα το μετανιώσουμε κάποια μέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πάντα, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε αυτή την ακρόαση. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. I Ίσως να ήταν πολύ πιο εύκολο να λύσουμε τα προβλήματα των χωρών αυτών παλαιότερα. Θυμάμαι κάποιες παλιές ε, ε, ε, τις που έγιναν με την συμφωνία του Παρισιού το 98-99 ήταν τότε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και εκτιμούμε πάρα πολύ τα όσα κάνατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωζώνη και ίσως και για τον κόσμο για έτσι μια γενική παγκόσμια λύση των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ. Next meeting is Monday, 7 p.m. in Strasbourg.